Άρα εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Ε, Ανακοινώσει του Προέδρου, σημείο 2. Όπως ξέρετε, το ΕΛΚ έχει μία συνάντηση τώρα στη Βιέννη, αν δεν κάνω λάθος. Και γι' αυτό τα μέλη από την πολιτική αυτή ομάδα δεν μπορούν να παρούνται στη σημερινή μας συνεδρίαση. Ένα κατάλογο τη αλληλογραφίας που έλειφθη μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνεται στου φακέλους των βουλευτών. οποίο θέλει να παρουσιαστεί κάποιο θέμα, είχε πραγματικέ πληροφορίε να ζητήσει από τη γραμματεία. Θα ήθελα να σα πω ότι η επόμενη μα συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση μα αυτή μάλλον θα περάσει στο web stream, Εκτό βέβαια το τμήμα και κλεισμένο των θερών τη συνεδρίαση. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο επόμενο θέμα. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των, του ρόλου των συντονιστών και εντολή για να λάβουν κάποιες αποφάσεις εξ ονόμου συνεδρίασης βάσει του άρθρου 192 του ιστορικού κονοσμού που λέει ότι οι συντονιστές μπορούν να προετοιμάσουν ε, πάνω σε αποφάσεις για την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την κατανομή των εκθέσεων στους ε, ε, αρμοδίους και επίσης θα μπορεί η Επιτροπή να αναθέσει την εντολή να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από τον, ε, τους συντονιστές εκτός από γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω η Επιτροπή Ήτρα να δώσει εντολή στους συντονιστές για να αποφασίσει τα εξής θέματα. Ακροάσεις, αντιπροσωπείες συμπεριλαμβανομένων και άλλων αντιπροσωπείων και μελέτες. Όσον αφορά τις αποφάσεις για τη ε, διαδικασία, τον ορισμό των εισηγητών, η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τις προτάσεις των συνοστές και θα τις επιβεβαιώνουμε, εάν δεν διαφωνεί κανένας. Αυτή είναι η πρότασή μου. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο συμφωνείτε. Έχει συζητηθεί και με του συντονιστέ αυτό. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Α περάσουμε τώρα στο θημείο 3. Έχουμε την κυρία Εύα Μπιόλινγκ, Υπουργό Εμπορίου τη Ιταλικής Κυβέρνηση, που εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου και θα μας παρουσιάσει τις επιτεύξεις της Ειδικής Προεδρίας στον τομέα της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής. Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω για μια φορά στην Επιτροπή μας, κύριε Υπουργέ ε, Εξωτερικού Εμπορίου της Συνδικής Κυβέρνησης. Έχει έρθει η στιγμή για τον απολογισμό, μια που λίγη προσεχώς η θητεία της Ειδικής ε, Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας ετέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας όπως ξέρει που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής θα είναι πια συνομοθέτης. Ε, τελευταία στην ε, Υπουργική Συνέλευση στην Γενέβη και η γραμματεία μας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Υπουργείου σας για να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και καλύτερη κατανόηση των αμοιβαίων θέσεών μας. Τώρα μας στα πλαίσια των θα προχωρήσουν οι σχέσεις της Επιτροπής εδώ με το Συμβούλιο και ελπίζω να υπάρχει πλήρης κατανόηση μεταξύ μας προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής δέχτηκα μία ε, η πρόσκληση για τις 12 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Εμπορίου και με τους συναδέλφους σας εκεί θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να εντείνουμε τις σχέσεις μας. Θα σας δώσω τώρα το λόγο για να μας κάνετε τον απολογισμό, όπως είπαμε, της Σουηδικής ε, Προεδρίας για το παρελθόν και για τις ευκαιρίες κατά που θα προσφέρει η συνθήκη της στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικά της εδώ Επιτροπής ειδικά και του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που επανακάμπτω εδώ στην Επιτροπή σας για να σας αναφέρω της, ε, τον απολογισμό της Ειδικής Προεδρίας στα θέματα εμπορικής πολιτικής. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σας αλλά και εσάς ε, για το νέο ρόλο που αναλαμβάνετε μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Γιατί η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα έχει ακόμη πιο εξέχοντα ρόλο σε θέματα εμπορικής πολιτικής από εδώ και πέρα, κάτι που είναι ευάρεστο και για την Προεδρία. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συνεργάστηκαν προωθώντα τη θέση Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και στην ανάπτυξη και σύσφυξη των εμπορικών τη σχέσεων. Με τη δική σα εμπειρία και την προστιθέμενη αξία που και στο μέλλον θα προσφέρετε στο θέμα του εμπορίου θα είναι πολύ χρήσιμα. Η Σουηδική Προεδρία επικεντρώθηκε κυρίω στα θέματα χρηματοπιστωτικής κρίση και τι επιπτώσει τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια ύφεση που είναι η βαθύτερη και ευρύτερη των τελευταίων γενεών. Και μάλιστα τα, οικονομικές προβλέψεις ευτυχώς ε, είναι πιο αισιόδοξες τελευταία και δείχνουν μια γενικότερη ανάκαμψη. Νομίζω ότι περάσαμε το χειρότερο τμήμα της κρίσης. Παρ' όλα αυτά η ανάκαμψη είναι ακόμη ευάλωτη και περισσότερο μας ανησυχεί η επιδείνωση στην αγορά εργασίας. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι πολλοί κίνδυνοι ελοχεύουν σε ό,τι αφορά την υψηλή ανεργία και τη συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού. Μία κατάσταση που ενισχύει την πίεση για περισσότερο προστατευτισμό και απομόνωση. Γι' αυτό μια υπεύθυνη στάση των παγκόσμιων εμπορικών εταίρων είναι επιθυμητή ήμουν την περασμένη εβδομάδα στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στη Γενέβη. Εκεί με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα ότι υπάρχει συνένεση για το σημαντικό ρόλο του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά μια ομαλή οικονομική ανάπτυξη και παγκόσμια οικονομική ε, μεγέθυνση και ανάκαμψη. Κάποια μέτρα προστατευτισμού χρησιμοποιήθηκαν, αλλά περισσότερο ε, ως αποτρεπτικά μέτρα και επιδιώχθηκε ιδιαίτερη διαφάνεια. Ω υπουργό Εμπορίου είχα ως προτεραιότητα να κάνω ό,τι μπορώ για να συμβάλλω στην διατήρηση του ανοίγματο της αγοράς αλλά και στην αποτροπή του προστατευτισμού. Στην περίοδο αυτή της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε και ηγετικό ρόλο αλλά και υποοικοδομητικό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και μάλιστα αντιστάθηκε στον πειρασμό να ενδώσει σε μέτρα προστατευτισμού. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί δώσαμε πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για αποφυγή προστατευτισμού. Σημειώσαμε και ένα σημαντικό βήμα πρόοδου ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση μετά το πρόγραμμα της Λισαβόνας. Και χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί το Συμβούλιο διατράνωσε τη δέσμευσή του για άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για προώθηση του εξωτερικού εμπορίου. Το ίδιο έγινε και στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού, όπως δείχνουν τα συμπεράσματα της 4ης Δεκεμβρίου. Επίσης, ε, παρακολουθούμε εκ του και τη στάση των εμπορικών μας εταίρων. Το πλαίσιο της ε, στρατηγικής ε, της εμπορικής αγοράς ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γι' αυτό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν το επιχειρησιακό περιβάλλον για τους ε, εξαγωγείς μας και τις αγορές στόχους, ώστε και οι εμπορικοί μας εταίροι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κρατούν ανοιχτές τις αγορές τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μια φιλόδοξη και ισόρροπη κατάληξη του DDA θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαβεβαίωση ε, κατά του προστατευτισμού. Γι' αυτό και είναι σημαντική η προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Μία πολυμερή συμφωνία θα μας δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ πιο στέρεο και ευνοϊκό από ό,τι στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε αμύωτη την πολιτική πίεση και να δώσουμε όθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία, κάτι που προϋποθέτει ενθάρρυνση και παρότριση των εμπορικών εταίρων μας να προσυπογράψουν πλήρως την DDA. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, επιμονή στη συζήτηση των θεμάτων που βρίσκονται επιτάπητος. Κάναμε πολλά βήματα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κατευθύνουμε προς σωστή κατεύθυνση την DDA. Και μάλιστα η διακήρυξη του G20 στο Pittsburgh ήταν σημαντικός στόχος και θα πρέπει μέχρι τα τέλη του 2010 να διεκπαιρεωθεί ο γύρος των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την πιο φιλόδοξη συμφωνία εμπορίου όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, οι διμερείς σχέσεις ε, ήταν ε, σημαντική προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ε, Δημοκρατία της Κορέας ήταν ανεπιφύλακτα ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, FTA, έχει σημαντικά ωφέλη για τους εισαγωγείς και εξαγωγείς, γιατί καταργούνται οι δασμοί και άλλοι εμπορικοί και δασμολογικοί φραγμοί. Επίσης, η εφαρμογή τη Ανατολική Εταιρική Σχέση ήταν σημαντική προτεραιότητα τη Σουηδική Προεδρία. Η πρόθεση τη σταθερότητα, τη σωστή διακυβέρνηση και τη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή είναι στρατηγική σημασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντική πρόοδο σημειώθηκε και πρόσφατα και μάλιστα συνεχίζονται οι συζητήσει για τη νέα συμφωνία σχεδίση με την Αρμενία και τη Γεωργία με στόχο τη διαπραγμάτευση ε, σημαντικών και εκτενών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Και η Ουκρανία είναι στενός εμπορικός μας και σημαντικός για την εμπορική για την ενεργειακή συγγνώμη, ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά, αλλά πολλούς δρόμους έχει ακόμη να διανυθεί. Και η Ρωσία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος και η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη εκτός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ τη προσχώρηση τη Ρωσία ε, στον ΠΟΕ, αρκεί φυσικά να επιληθούν τα εκκρεμή εμπορικά ζητήματα. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στι διαπραγματεύσει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία. Επαναλαμβάνονται οι διαπραγματεύσει μετά από μια σύντομη διακοπή στι αρχέ του χρόνου. Η διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία ε, προώθησε σημαντικά τι διαπραγματεύσει για τη νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Σε ό,τι αφορά την Νοτιοανατολική Ασία, Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε τις διμερείς διαπραγματεύσεις με χώρες του ΑΣΕΑΝ και θα χαράξουμε το δρόμο για μελλοντικές περιφερειακές συμφωνίες. Έτσι θα υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας στόχο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού μας χάρη στην ενισχυμένη πρόσβαση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι διαπραγματεύσεις συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το Περού και την Κολομβία βρίσκονται σε καλό δρόμο και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να προαγάγει την διαδικασία αυτή για τη σύναψη συμφωνίας, ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με όλη την περιοχή των Άνδεων. Επίσης, οι συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική βρίσκονται σε καλό δρόμο, αλλά οι ατυχείς εξελίξεις στην Ονδούρα μας ε, υποχρέωσαν να αναστείλουμε τις διαπραγματεύσεις. Το θέμα της Ονδούρας θα πρέπει να επιληθεί πριν συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, για να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ονδούρα. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στις διαπραγματεύσεις ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με τον Καναδά. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένας ε, επιτυχής γύρος και ε, το μέλλον είναι βίωνο. Επίσης θα, θα συνάψουμε το και τη Μαδαγασκάρη, το Ζιμπάμπουε, τη Γουινέα συμφωνίες και μάλιστα το, Φθινόπορο το διοργανώσαμε το πρώτο διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Εκεί συζητήσαμε την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα νομοθετικά σε τομείς όπως η σήμανση, η ανατεχνολογία και η ενεργειακή αποδοτικότητα, προκειμένου να εθετήσουμε κάποιες συμβατές και συγκλίνουσες προσεγγίσεις για κανονιστικά θέματα. Επίσης, θα ξεκινήσουμε ένα νέο διάλογο καινοτομίας για να τονώσουμε την παραγωγικότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την οικονομική μεγέθυνση. Η 8η Υπουργική Διάσκεψη της Euromed έγινε χθε στις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί συμφώνησαν σε ένα οδικό χάρτη μετά το 2010 που διορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και για την ε, αποκατάσταση μιας ευρύς ε, ζώνης, ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην Ευρωμεσογειακή Λεκάνη. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι περιορίζεται η γραφειοκρατία στην περιοχή της ε, Euromed και μάλιστα χάρη στην ε, περικοπή τη γραφειοκρατίας θα μειωθεί και το κόστο των διασυνοριακών συναλλαγών. Σημαντικό βήμα αυτό στη συρρήκνωση τη γραφειοκρατία, ένα στόχο που θα ε, επιδιωχθεί και στο μέλλον. Γιατί οι λιγότερες γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες και διατυπώσει μειώνουν το κίνδυνο τη διαφορά. διαφθοράς και στην καταπολέμηση τη διαφθορά χρειαζόμαστε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Και μάλιστα η στη συνέλευση των ε, συμβολωμένων μερών στην Τόχα αποφασίστηκε ένας μηχανισμός ε, ε, επιτήρησης για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Κάτι που είναι μοναδική ευκαιρία για μας, γιατί θα βοηθήσουμε, θα, θα οι χώρες για την αποτελεσματική και εύρυθμη εφαρμογή της σύμβασης. Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν είχαν παραμείνει αμύωτες και επίμονες οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική πρόοδο συνιστά και η διευθέτηση ε, κάποιων εκκρεμών διαφορών, όπως είναι η συμφωνία με τη Βραζιλία σε ό,τι αφορά κάποια εκκρεμή ζητήματα που έμειναν από τι διευρύνσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε σημαντικέ διασκέψει κοινωνική με την Νότια Αφρική, τη Βραζιλία, τι Ηνωμένε Πολιτείε, Ινδία, Ρωσία, Κίνα και Ουκρανία. Θα ήθελα να τονίσω και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Την εταιρική ευθύνη και μάλιστα μια επιτυχής ε, συνδιάσκεψη για το θέμα αυτό έγινε τον Νοέμβριο στην Στοκχόλμη. Και αναφερθήκαμε στο ρόλο των κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τα, ανθρώπινα δικαιώματα και την εξασφάλιση της ευημερία των επιχειρήσεων αλλά και, τον και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα αυτό αναφέρεται και στα συμπεράσματα της 8 Η Δεκεμβρίου του Συμβουλίου. Η έκβαση της συνδιάσκεψης ε, συνοψίζεται σε μία δήλωση που θα σας δώσω στο τέλος της συνεδρίασης μαζί με την Ισπανική Προεδρία. Γιατί τώρα μεταδίδουμε τη σκητάλη στην Ισπανία, την επόμενη Προεδρία που θα προωθήσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το πλαίσιο αυτό, αλλά και την έμπρακτη εφαρμογή του. Σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία κατά της παραποίησης, έχουν γίνει μέχρι στιγμής δύο γύροι διαπραγματεύσεων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, εφαρμογής πρακτικών και ενίσχυσης πρακτικών, θεσμικά ζητήματα, ποινικέ κυρώσεις, το ψηφιακό περιβάλλον και τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω πρόοδο κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και ευχόμαστε για την αίσια κατάληξη των διαπραγματεύσεων κατά το 2010. Η εμπορική πολιτική μπορεί και ε, οφείλει να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Η συνοχή μεταξύ της εμπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής είναι σημαντική για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικός εταίρος των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Η σχετική πολιτική ανάπτυξη έρχεται τον Νοέμβριο. Τα συμπεράσματα γίνουν μια σειρά προτεραιοτήτων για την, ε, το εμπόριο και την ανάπτυξη, όπω είναι βελτιωμένη και αποτελεσματική πρόσβαση αναπτυσσομένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ελεκτρικό σωπόδιο, η προώθηση τη υφόρου ε, ανάπτυξη και μέθοδη καλύτερη χρήση των διεθνών δικαιωμάτων πνευματική ε, ιδιοκτησία καινοτομία και ανάπτυξη. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να βασίσουμε τη μελλονική μας εργασία στα πιο κέρια θέματα μεταξύ ανάπτυξης και εμπορίου. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα της ανάπτυξης θα είναι κάτι που θα πρέπει να είναι πάντα κατά νου μας ε, όταν εξετάζουμε την ε, εμπορική πολιτική. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την εμπορική πολιτική είναι οι κλιματολογικέ αλλαγέ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλε τι δυνατότητε που προσφέρει το εξωτερικό εμπόδιο για να καταπολεμήσουμε τι ε, αλλαγέ αυτέ. Καταβλήθησαν προσπάθειε να προωθηθούν οι συζητήσει για την απελευθέρωση του εμπορίου φιλικών προ το περιβάλλον ε, εμπορευμάτων μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλό να το πετύχουμε αυτό και τώρα ενώ ώψη διαπραγματεύσεων για τι κλιματολογικέ αλλαγέ τονίζουμε τη σημασία τη ισχυρή προστασία και ενδυνάμωση των προσπαθειών μας για να ενισχύσουμε την καινοτομία και επενδύσεις στην, ε, ε, στις τεχνολογίε. τεχνολογίες. Η διάσκεψη στην Στοκχόλμη για, την, ε, για το εμπόριο και την τυποποίηση στον αντισυκό τομέα έγινε στο Στοχόλμη τον Νοέμβριο και πιστεύουμε ότι οι κλιματολογικές αλλαγέ θα είναι ένα θέμα που θα επανέρχεται συνεχώς στην ε, ατζέντα της εμπορικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Επίσης ε, ξεκίνησα μία συζήτηση για το μέλλον του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Θα πρέπει να ανταποκριθεί στις σημαντικότητε αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στη διεθνή οικονομία Όπω σας είδαμε τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο δρούν οι επιχειρήσει έχει αλλάξει σημαντικά. Το εμπόριο σήμερα μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι δραστηριότητα μεταξύ δύο κρατών. Συνήθως είναι μία διαπραγμάτευση μεταξύ επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι εξαρτώνται σήμερα από τις ε, διεθνείς ε, ε, αλυσίδες ε, συναλλαγών και τη διεθνή παραγωγή. Θα μπορέσουμε νομίζω να έχουμε μία να σας πω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση στην επίσημη Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου το Σεπτέμβριο. Η 7η Σύνοδος που επίσης είχε την δυνατότητα να συζητήσει γενικά το θέμα του διεθνού εμπορικού συστήματο. Όσο πάει και περισσότερο αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρχει νέα σκέψη, νέα μέθοδο πολιτική. και ελπίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή με το εξωτερικό εμπόριο. Πιστεύω ότι μόνο με μια ανοιχτή, ενεργή, συνεπή και αηφόρο εμπορική πολιτική θα μπορέσουμε να πετύχουμε ανάπτυξη και ευμανία προ όφελο των πολιτών μα. Προσβλέπω λοιπόν στην περαιτέρω συνεργασία με το Κοινοβούλιο στα τόσο σημαντικά αυτά θέματα του του θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την προσοχή σας και να σας πω ότι με χαρά θα ακούσω τα δικά σας σχόλια και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχόλια και στις ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Now let's go. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να δούμε τώρα ποιος ε, έχει να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις. Εγώ εκμεταλλόμενος το προνόμιο του πρόεδρου, θα σα υποβάλω την πρώτη ερώτηση. Είπατε εισαγωγικά στην, για την ε, Σουηδική Προεδρία. Είχατε πει ότι ο γύρο τη Δόχα ήταν ε, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη προτεραιότητα τη ε, σα. Δυστυχώ όμω δεν νομίζω ότι είχαμε πραγματική πρόοδο. Πρόσφατα ήμασταν στη Γενέβη και διαφάνηξε κάθαρα ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για να καταλήξουμε σε μια επιτυχή ενδεχομένω ολοκλήρωση του γύρου της Δόχα. Κατά τη γνώμη σας, γιατί υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις. Και πιστεύετε ότι να ολοκληρωθεί ο γύρος αυτός μέχρι τα τέλη του έτους, του επόμενου έτους. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάρτιν Κάζακ της ε, ομάδας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω για όλες τις ε, προσπάθειες, ε, τις δικές σας προσωπικά και της ε, Σουηδικής Προεδρίας για να προχωρήσουμε σε θέματα καυτά για την εφαρμογή της κοινή εμπορικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες διαφορές αντίληψης ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών και των ενδιαφερομένων για αυτά τα θέματα. Να θυμίσω και αυτό το οποίο είχατε πει τον Σεπτέμβριο στην τελευταία μας ακρόαση για τη Συμφωνία Ελευθέρων Ανταλλαγών με την Νότια Κορέα. Είχατε πει ότι πρόκειται για μια τεράστια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η συμφωνία Είχατε πει λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία ήταν πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη ΣΑΜΠ και τη Volvo, ε, αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης με 400, 400 άτομα τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους. Είχατε πει ότι αυτό δεν ήταν ε, πρόβλημα υπήρχε μία δυνατότητα ε, να μεταφερθούν ε, ε, αυτοί οι εργαζόμενοι να μετατεθούν σε άλλες επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας, καινοτομίας κλπ. Μετά από τέσσερις μήνες εσείς πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια καλή και συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάντοτε διαφορές εσείς ε, διαπιστώνετε να υπάρχουν κάποια μηνύματα από την Κομισιόν για να ε, ε, χρησιμοποιήσει τη ρήτρα διασφάλισης πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεύτερη ερώτηση, σχέσεις με την Ουκρανία. Ξέρετε ότι η Ουκρανία σταμάτησε την είσοδο του, Μαυροβονίου στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ε, για λόγους άγνωστους, φαντάζομαι κατόπιν πιέσεως της Σερβίας. Εσείς θα, θα, παίξετε διαμεσολαβητικό ρόλο για να λυθεί το πρόβλημα. Τρίτο, για την Ρωσία η Ρωσία θα προχωρήσει σε τελωνιακή ένωση με το Καζακστάν και την Λευκορωσία, πράγμα που θα καθυστερήσει την είσοδο της Ρωσίας στην ΠΟΕ. Λοιπόν, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα είμαστε στη δέκατη μέρα από τη θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να διευκρινίσουμε ποιος είναι ο ρόλος και η εντολή των τριών θεσμικών οργάνων για την εφαρμογή αυτής της συνθήκης. Πολλοί ζήτησαν το λόγο να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Ο κύριος Μάικλ Φάρελ από την Άλντε επίσης. Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας συγχαρώ και σας και τη Σουηδική Προεδρία για την τόσο επιτυχή σας εργασία των τελευταίων ημών. Για εμάς τους βουλευτές ε, με την 1η Δεκεμβρίου και την θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα Λισαβόνας ε, είδαμε να περνάει ένα σημαντικό, μια σημαντική ημερομηνία και θέλω να σα χαρώ ω τη αντιπροσωπεία στη Γενέβη τις ε, περισμένες αυτές ημέρα τη Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου μου δημιουργήθηκε μια ερώτηση από όσα είπε και ο Πασκάρ Λαμή και η Επίτροπος Μάνιο Φισερμπέλ δημιουργήθηκε εντύπωση ότι τους επόμενους τρεις με πέντε μήνες θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση για να προωθηθεί ο γύρος της Δόχα για να μπορέσει να καταλήξει κάπου και να καταβάλει κάθε προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί η πρόοδος όπως το τόνισε και ο πρόεδρος Μορέρα. Έξω και η ερώτησή μου. Στο ψήφισμά της για το γύρο της Δόχα, η πολιτική μου ομάδα ανέφερε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει, να ε, παρουσιαστεί σαν μια γέφυρα μεταξύ των ΗΠΑ αφενός και των άλλων χωρών αφετέρου, εσείς φαντάζεστε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντολή για μια τέταρτη δευτερότητα γεφύρωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Ο Μπέρν Λάγκ έχει το λόγο, σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θα σα ευχαριστήσω για όσα μα είπατε. Θα ήθελα να υποβάλω ε, ερωτήσεις για δύο θέματα. Τονίσατε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να προωθήσει και την ανάπτυξη. Και αυτό βέβαια εν ώψη του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει συμφωνία με τις χώρες των Άδεων. Δεν ξέρω. Εσείς είπατε ότι είναι καλό αυτό. Είναι πράγματι όμως καλό. Είναι αληθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το δύο χωρών των Άδεων... που παραμένουν στις διαπραγματεύσεις εν αντιθέσει προς τη ΣΥΠΑ ζητάει μακρύτερη περίοδο προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα. γιατί αυτή τη στιγμή το 70% αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων είναι τα λεγόμενα no-name και γιατί εσείς ε, θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια προστασίας. Δηλαδή η ΕΠΑ ζητάνε μόνο 10, η Ευρωπαϊκή Ένωση 15 χρόνια. Μετά, τι γίνεται όσον αφορά με την προστασία των δικαιώματων επί της γης, μικροπαραγωγών και ε, χωριών. Και τρίτον, τι γίνεται με τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως στην Κολομβία. Η Κολομβία είναι γνωστό. Είναι εκείνη η χώρα στην οποία τα συνδικαλιστικά δικαιώματα καταπαντούνται. Το 70% όλων των βίων πράξεων κατά συνδικαλιστών λαμβάνουν χώρα στην Κολομβία. Και εγώ δεν έχω καμία κανένα όταν και το Κογκρέσο των ΗΠΑ και η Βουλή στον Καναδά και στην Νορβηγία επίσης. Το Συμβούλιο, ε, μάλλον εκείνες, αυτές οι χώρες ε, διακόπτουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το κάνει για να περιμένει να γίνουν σεβαστά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στις χώρες αυτές. Μήπως θα πρέπει να ακολουθηθεί και εδώ μια διαφορετική άγουσα. Και κατόπιν αναφέρω και σε αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, κύριε Πρόεδρε. Τι αποφάσισε συγκεκριμένα το Συμβούλιο, ποια είναι τα μέτρα που θα εφαρμόσει για να πραγματοποιηθεί, να ακολουθηθεί η συνθήκη της Αβώνης. Πώς θα εμπλέξει στο μέλλον το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο σε διαπραγματεύσεις για εντολές και επίσης πώς θα εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο ισότιμα στην Επιτροπή 133 όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων αυτών με τρίτες χώρες ενώ πάντα. Και επίσης θα υπάρχουν παρατηρητές στις διαπραγματεύσεις όπως και το Συμβούλιο στέλνει παρατηρητές σε κάποιες διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, Πώς θα δώσετε πνοή και ζωή στη Λισαβόνα. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Ντέβιτ Μάρτιν, ε, πάλι από το δύο κόμμα και Δημοκράτες. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα, για, ιδιαίτερα για την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κολομβία. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει στις διαπραγματεύσεις συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου να έχουμε ε, ρήτρες τύπου TRIPS TRIPS-SYN Και ήταν σαφές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ρήτρα ρήτρα TRIPS-SYN είναι απαράδεκτο να περιλαμβάνεται σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Ε, είστε τυχεροί που η συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ επί της Προεδρίας σας. Είχατε μέχρι στιγμής διεξοδική συζήτηση στο Συμβούλιο για το νέο ρόλο που θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη θέση εφαρμογή της Σύνθηκης Λισαβόνας και πώς θα λειτουργήσει η νέα δυναμική στις σχέσεις μας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μας στέλνετε όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Η δική μας γνώμη είναι θα είμαστε σαφώς πιο αναμειγμένοι. Εσείς τι πιστεύετε, θα συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της διαπραγματευτικής εντολής για τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Πώς θα μας ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις, ώστε στο τέλος της διαδικασίας αυτής να μην υπάρχει αποσύνδεση και απογοήτευση μεταξύ των δικών μας προσδοκιών για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και του τελικού αποτελέσματος. Σε ό,τι αφορά θέματα δασμολογικών προσαρμογών, θα συζητήσουμε αργότερα συμφωνίες με προμηθευτέ μπανάνας. Η δική μου γνώμη είναι κατηγορηματική ότι τέτοιε συμφωνίε θα πρέπει να επικυρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι χρειάζεται και αυτό το θέμα στην απόφαση. Τι λέει η δική σα νομική υπηρεσία. Για ένα διαφορετικό θέμα τώρα, την Κορέα. Τη συζητήσαμε και στο παρελθόν, α μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Πάντω, όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά κυρίω εσεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καταφέρατε να περάσετε το μήνυμα για τα ωφέλη που θα έχει η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κορέα. Οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν σε θέματα αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν νομίζω ότι θα βγει τόσο χαμένη όσο προτάθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία. Άλλωστε υπάρχουν πολύ περισσότερα ωφέλη. Και σίγουρα θα κερδίσουμε πολλά από το γεωργικό κλάδο. Κάτι που δεν είναι εύκολο θα κερδίσουμε στα φαρμακευτικά, θα κερδίσουμε στη γεωργία, στα, στους ίνους κοινοπνευματόδη από αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Επίσης θα κατοχυρώσουμε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε θέματα τραπεζικά και υπηρεσιών θα αποκομίσουμε πολλά ωφέλη σε θέματα πρόσβαση αγοράς. Είναι τεράστια τα προτερήματα αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ε, η μελέτη της Στοκόλμης λέει ότι θα στοιχήσει 91,1 δις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και όταν ακούτε τις συζητήσεις ε, αποκομίστε την εντύπωση ότι εμείς όλο υποχωρήσεις κάναμε προς την Κορέα για τη συμφωνία αυτή, ενώ το αντίθετο συμβαίνει. Ο κύριος Καντέρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για τον απολογισμό που κάνατε. Σχετικά με μερικά πράγματα που είπατε, σχετικά με τη συνοχή. Θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι πολλά πράγματα μας ε, χωρίζουν. Για την Κολομβία, εσείς εκφράσατε ικανοποίηση που συνεχίζονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Κολομβίας και Περού αλλά για μας ε, στην ε, ομάδα των σοσιαλιστών δημοκρατών ε, και κατά τα λεγόμενα των κολομβιανών συνδικαλιστών ήταν απαράδεκτο να συναυθεί μια συμφωνία με την Κολομβία σήμερα. Καταπατούνται συνδικαλιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα και πραγματικά η η Ευρωπαϊκή Ένωση αειδός των ε, με ομικρονιώτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν μπορεί να υπογράψει συμφωνία με την Κολομβία. Το ίδιο ισχύει και για το Περού και για την ε, Σαβιλάνκα. Και τώρα για να είμαι συνεπής για την Νότια Κορέα, ορισμένα πράγματα μας χωρίζουν τους μεν από τους δε, αλλά η συνοχή είναι κάτι και η συνέπεια είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας καίει στην ομάδα μου. πέρα από τα θέματα γεωργίας, βιοτεχνίας ε, ε, κλπ. θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και το θέμα της βιομηχανίας. Η βιομηχανική πολιτική και οι εμπορικές συμφωνίες δεν είναι άσχετες μεταξύ τους. Οι πολίτες ε, ενδιαφέρονται άμεσα για όλα αυτά. για τις συμφωνίες με την Αφρική. Μερικοί από εμά πήγαμε στην ε, Λουάντα της προάλλες για τη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Και καμιά αφρικανική χώρα, από ό,τι ακούσαμε εκεί πέρα, δεν είναι ευχαριστημένη με τις διμερείς συμφωνίες. Η ακτή του ελεφαντόδοντος δεν έχει καμία όρεξη δεν να προχωρήσει παραπέρα. Υπάρχει ένα φόρουμ που ψηλολειτουργεί, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι εντελώς αποτυχία. Θέλω να ξέρω τι λέει το Συμβούλιο για όλα αυτά. Εμπορική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική, θέλω να ξέρω τη θέση σας. Διότι εντάξει λέμε εμπορική πολιτική πρέπει να βοηθάει την αναπτυξιακή πολιτική, αλλά άμα δεν βάζουμε και τα μέσα στη διάθεσή της για να πετύχει, τι γίνεται. Ξέρω θα μου πείτε εγώ δεν είμαι υπεύθυνη. Διότι εντάξει εμπορική πολιτική, αλλά υποχωρώντα σε θέματα παιδείας και άλλα δεν βοηθούμε την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Θέλω να ξέρω λοιπόν στις νέες συμφωνίες που θα υπογραφούν ποια είναι η θέση σας μας, για αυτήν την αντίφαση, δηλαδή γενεοδορία από τη ΜΕΑ αλλά κανένα μέσο για να την πετύχουμε. Ευχαριστώ κύριε. Καδέρο, κύριος όλους από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για τις σχέσεις ε, ανάπτυξης και διεθνούς εμπορίου. Και μάλιστα αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε την κατάσταση του διεθνούς εμπορίου μεσούς της κρίσης. Γιατί η κρίση διαρκεί και σίγουρα οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι πλέον ευάλωτες απέναντι σε αυτή τη χρηματοπιστωτική κρίση. Έχω μια ερώτηση σχετική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβαμε υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, ότι η ανάπτυξη και το διεθνές εμπόριο ήταν ανέκαθεν ε, προτεραιότητες της ε, Προεδρίας σας. Εμείς, η Γκουέ, αλλά και εγώ προσωπικά, Έχω πολλές αφιβολίες για το κατά πόσο ήταν θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα μιας ε, ευόδοσης των διαπραγματεύσεων της Ντόχας για την συμφωνία σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους. Μπορείτε να μας αναπτύξετε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα. Πώς συνδέεται δηλαδή τα αποτελέσματα του τρέχοντος γύρου με την ε, δεδηλωμένη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη συνάφεια ανάπτυξης και εμπορίου. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε διεθνείς συμφωνίες ε, όπως για το κακάο και το καφέ που είναι ακόμη πιο σημαντικές εν μέσω αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Και φυσικά να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των τρίτων χωρών με τις οποίες έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Αναφέρθηκατε και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς σκοπεύετε απτά και συγκεκριμένα να αντιμετωπίσετε το διεθνές εμπόριο ως μέσω των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Γιατί το Κοινοβούλιο, χάρη στην εκτεταμένη συναπόφαση, θα είναι πολύ πιο ε, εφοδιασμένο να αντιμετωπίσει τις ε, μελλοντικέ προκλήσεις και γι' αυτό θα πρέπει και η Προεδρία να μας δώσει πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για την έμπρακτη εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης Λισαβόνας και την σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Ή πώς σκοπεύετε εσείς και η Κομισιόν να εφαρμόσετε ή να λάβετε υπόψη τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου στα πλαίσια της συναπόφασης. Αναφέρθηκαν ήδη συμφωνίες για τις μπανάνες. αν ολοκληρωθεί ο στόχος, ε, αν ολοκληρωθεί ο γύρος της τι θα γίνει σε σχέση με τις μπανάνες τι γίνεται ε, με, το μηχανισμό της του ΠΟΕ για την επίλυση των διαφορών. Μήπως ε, θα υπερφορτωθεί αυτό το, το πάνελ με διάφορες τέτοιες ε, εκρεμείς διαφορές εφόσον δεν ε, ολοκληρωθεί ο κύριος της Ντόχα. Η Μαρία Μουνής από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. A la presidencia sueca. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της αηφόρου ανάπτυξης στη συμφωνία με την Κολομβία που θα επιτρέψει να ανοίξει ένας διάλογος και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έστω και αν είναι μια μερική συμφωνία με την Κολομβία και όχι μια συνολική συμφωνία με όλη την περιοχή, αυτό θα επιτρέψει να ανοίξει μια, ε, μια πόρτα επιρροής ε, για την, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να ξεκινήσει και μια παρέμβαση της ε, ΔΟΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα για τις μπανάνες θα ήθελα να ολοκληρώνουμε τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό διότι αυτό θα έλυνε όλες τις ε, προηγούμενες ε, συγκρούσεις και θα απολευθέρωνε και τη δυνατότητα υπογραφής όλων των υπολείπων εκκρεμών διμερών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Δεν έχει άλλο το λόγο. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην επισκέπτριά μας να απαντήσει. Παρακαλώ. Εγώ σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Από ό,τι κατάλαβα έχω 7 λεπτά για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις αυτές, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Θα αρχίσω με το πιο γενικό ερώτημα του Προέδρου για το κύριο της Ντοχά. Δεν υπάρχει πρόοδος. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει και αποτυχία. Είμαι πολύ ε, περήφανη που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε και θέλει να ολοκληρωθεί ο γύρο ε, της Δοχά. Είχαμε μια συνάντηση πριν αρχίσει η συνάντηση ΠΟΕ και υπάρχει έντονη υποστήριξη από τα κρατημένα για να προωθήσουμε την ε, τελειοποίηση τη γύρω τη Δοχά το 2010. Υπάρχουν και ορισμένα βέβαια εταίροι που δεν είναι ακόμα προετοιμασμένη για την ε, τελική διαπραγμάτευση. Πρέπει είπα να έχουν την σαφή εντολή. Αυτό μας λείπει σήμερα. Και πριν να το πετύχουμε, δεν θα δίνουμε ούτε την Κίνα, ούτε την Βραζιλία, ούτε την Ιδία να δείξουν κάποια ευελιξία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να κατονομάζουμε και ντροπιάζουμε name ναι, and shame εδώ. Αυτό δεν θα μας βοηθήσει. Καλύτερα είναι να φροντίσουμε να δούμε πώς θα μπορούμε να διευκολύνουμε τις χώρες αυτές να επανέλθουμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με σαφή εντολή να δείξουμε ευελιξία, να τους υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα γύρο αναπτυξιακό και το ε, Διατλαντικό Συμβούλιο Οικονομικών θα πρέπει να βοηθήσει εδώ. Χρειαζόμαστε όλους τους διαφορετικούς εταίρους να συνενεθούν για να προχωρήσει ο γύρω Σιλόχα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη προτεραιότητα. Γιατί αυτό θα αποστείλα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ιδίως μετά από αυτή την οικονομική κρίση που ε, ζήσαμε, γιατί πρέπει να διευκολύνουμε το διεθνές εμπόριο, αυτό θα βοηθήσει πολύ όλες τις χώρες. Και θέλω να φέρω και κάτι πολύ το θετικό στις που έχει τώρα στη Γενέβη, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες κατοφλίου τουλάχιστον, ε, πρόσφατα ε, βιομηχανοποιημένες, τόνισαν πόσο το χρειαζόμαστε όλοι. Το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ αυτό. Άκουσα κάποια σχόλια για τη συμφωνία με την Νότιο Κορέα και τη σημασία της και είπα ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα να μπορέσουμε να τελειοποιήσουμε ιδίως στη εποχή οικονομικής κρίσης. Και θα ήθελα να διορθώσω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι πρόβλημα στη Σουηδία. Αυτή η 4.700 ανεργοί, τεράστιο είναι το πρόβλημα. Αλλά από την άλλη μεριά το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τα χρήματα των φορολογουμένων και επιδοτήσεις στη βιομηχανία. Είπαμε ότι θα πρέπει να προσφέρουμε άλλες δυνατότητες για να δημιουργηθούν και άλλες ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς. Γιατί υπάρχουν, ε, παραδείγματο χάρη, δυνατότητε στον ε, τομέα έρευνα και ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο να πούμε ότι πρόκειται για ένα διορθωτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δεν σχετίζεται καθόλου με την Νότιο Κορέα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πολλοί άλλοι Αναφερθήκανε στην αυτοβιοικονομία στην Νότιο Κορέα. Άκουσαν τον Μάρτιν Ντέβιτ από τους συζητητές και δημοκράτες και άλλου. Θα έπρεπε ίσω να προχωρήσουμε λίγο παρατέρα στι λεπτομέρειε. για την Νότιο Κορέα. αναφέρθηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους μη Ευρωπαίους ε, εμπορικούς εταίρους. Είχαμε μια αύξηση 10% μεταξύ 2003 και 2007 και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό της διεθνούς ε, ατζέντα της Ευρώπης και ένα σημαντικό μήνυμα ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και με άλλες διαπραγματεύσεις. θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς όπως παρουσιάστηκε πολύ ωραία και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω 100% με αυτό που ελέγχθη σχετικά. Ότι συγκεντρώθηκε η προσοχή στην αυτοκινητοβιομηχανία παρόλο που συμπεριλαμβάνουν και πάρα πάρα πολλοί άλλοι τομείς σημαντικοί για μα. Και ότι αυτό πρόκειται για μία συμφωνία που θα οδηγήσει σε όφελος και τα δύο μέλη. Μετά, όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης, υπαναχώρηση και διασφάλιση, όπως συζητήθηκε το φθινόπωρο. We should reflect that uh, the fact that Korea already allows duty drawback. Ε, υπήρχε ένας ε, συμβασμός ότι η Κορέα επέτρεψε κάποια επαναχώρηση και ότι υπάρχει στο, θα υπάρχει στο μέλλον ε, περισσότερη συνεννόηση και με την Κίνα για το θέμα αυτό. Αυτό οδηγεί σε μηχανισμούς που αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Κάποιο είπε ότι οι προσπάθειέ μα δεν είναι αποτελεσματικέ. Εγώ διαφωνώ. Θα ήθελα να σα πω ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού θα πρέπει να βοηθεί από εμά ανεξάρτητα. Και θα ήθελα να σας πω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν λάβει τη δέσμευση να προσπαθήσουν η εφαρμογή να είναι αποτελεσματική. Και επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειες μέσα στα πλαίσια των κανόνων FTA για τη λεγόμενη εσωτερική επεξεργασία. Θα σταματήσω εδώ νομίζω για την αυτοβιομηχανία. Then Σχέσεις με την Ουκρανία τώρα. και την προσπάθειά της να κόψει το δρόμο του Μαυροβουνίου. Στην Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Γενέβη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε στεναρά την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στον ΠΟΕ και διευκρίνησε ότι το αίτημα της Ουκρανίας για το Μαυροβούνιο είναι απαράδεκτο σε αυτή τη φάση. Σχέσεις με τη Ρωσία. Τελωνιακή Ένωση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν. Όπως είπα και στην ομιλία μου, είναι ύψητη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Με τις ίδιες όμως προϋποθέσεις που ισχύουν και για τα άλλα μέλη του ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που λαμβάνουμε για την Τελωνιακή Ένωση με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν, είναι σημαντικό να είναι σαφή αυτά τα μηνύματα ότι η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και αυτής της χώρας. Στη Στοκόλμη πάντως, ε, στην πρόσφατη διάσκεψη που είχαμε με Ρώσους ομολόγους, λάβαμε σαφές μήνυμα για την προσήλωση της Ρωσίας στο θέμα της ένταξής της στον ΠΟΕ. Και μάλιστα ως ένα κράτος. Then uh, we had uh, uh, ερώτηση από τον Μπεν Λάγκε των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τα θέματα των TRIPS και τα αναπτυξιακά ζητήματα. αλλά και για την Κολομβία. Το θέμα της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Κολομβία το επισήμαναν πολύ. Ο Μπέρντ Λάγκε ρώτησε και για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ερωτήματα άλλωστε που ήταν κοινά σε πολλές ε, παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω με τα τρίψη. γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, τη δήλωση των TRIPS και τα θέματα δημόσιας υγείας. Πρόθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είδε είναι να υπονομεύσει την ελαστικότητα των TRIPS με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες. Η ελαστικότητα είναι απαραίτητη στην περίπτωση αυτή για να εξασφαλιστεί και η γενικότερη ισορροπία της συμφωνίας. Βέβαια δεν αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση διμερώς με τους εταίρους της ε, να βρει κάποιες λύσεις που θα συμπληρώνουν ε, τα TRIPS, αν κρυθεί σκόπιμο. Θα γίνει όμως μια κατά ανάλυση όλων αυτών των περιπτώσεων, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της ε, δεδομένης χώρας. Για το θέμα της Κολομβίας, δυστυχώς συνεχίζεται η βία και η καταστολή, η καταπίεση κατά των συνδικαλιστών στην Κολομβία, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αποτελεί ακρογωνίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας με την Κολομβία και μάλιστα ήδη έχουμε δώσει έμφαση στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συνομιλίες μας με την Κολομβία. Πάντως, είναι σημαντικό να δίνουμε, παρουσία στις να δίνουμε το παρόν στις χώρες αυτές και να διευκολύνουμε τις εμπορικές συναλλαγές μαζί τους, γιατί με τέτοιες ενισχυμένες ε, σχέσεις και συναλλαγές μπορούμε να επηρεάσουμε ε, χάρη στις ε, επιχειρήσεις μας και να δώσουμε το παράδειγμα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, να τονίσουμε την ανάγκη της εταιρική και κοινωνικής ευθύνης για να δείξουμε και εμείς πως εφαρμόζουμε εμπράκτος τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργώντα μια άμυλα και προς τις χώρες αυτές. Επόμενη ερώτηση αφορούσε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος για τη θέση ισχύ της νέας συνθήκης. Το είπα και στην ομιλία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρη στην εκτεταμένη εφαρμογή της διαδικασίας συναπόφασης, οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου θα ενισχυθούν. Γι' αυτό θα πρέπει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζονται στενά και με επικοδομητικό τρόπο για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας. Θα γίνουν συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τη συγκεκριμενοποίηση της συνεργασίας μεταξύ μας. Για παράδειγμα, πώς θα ενημερώνεται το, το Κοινοβούλιο για διάφορα θέματα. Ήδη ξεκίνησε η σχετική συζήτηση Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης ε, και το περιεχόμενο της ενημέρωσης και την έκταση της ενημέρωσης, το Κοινοβούλιο θα δικαιούται την ίδια ενημέρωση με το Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 207. Τώρα, πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε μεταξύ τους στα δύο θεσμικά όργανα. Πάντως, και αυτό το συζητήσαμε στο πρωινό που είχαμε με τους ευρωβουλευτέ στη Γενέβη. Για το... Θα φροντίσουμε να εφαρμοστεί εμπράκτο αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Το Κοινοβούλιο και ο αρμόδιος ε, Υπουργός, ο ε, ε, αρμόδιος Επίτροπος Εμπορίου καθώς και το Συμβούλιο ε, θα πρέπει να συζητήσουν ε, για το πώς θα δώσουν σάρκα και οσά αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να γίνουν σχετικά γρήγορα και με ομαλό και εύρυθμο τρόπο. Πάντως θα πρέπει κατεπηγόντως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να βρουν τους καλύτερους τρόπους συνεργασίας για να μην δημιουργηθεί καμία καθυστέρηση στη συναπόφαση. Uh, uh, Maria Muniz Η Μαρία Μουνής έθεσε ένα ερώτημα για τις μπανάνες. Συμφωνώ ότι είναι σημαντική μια συμφωνία για τις μπανάνες. και θα διευκολύνει και την ε, διεκπαιρέωση του γύρου της Δόχας. Βέβαια το θέμα αυτό είναι πολύ σύνθετο, οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί, γιατί έχουμε μπανανοπαραγωγούς στη Λατινική Αμερική, στις χώρες ΑΚΕ, αλλά και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η διαφορά της μπανάνας καλά κρατεί εδώ και 50 χρόνια περίπου στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Πάντως στη Γενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοντεύει να βρει συμφωνία με τα συμβαλόμενα μέρη και αισιοδοξούμε ότι η συμφωνία αυτή θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Αυτά για τις μπανάνες προς το παρόν. Τέθηκε και μία ερώτηση για τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, EPA. about the Όπως και το Σεπτέμβριο, η Σουηδική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στις συμφωνίες αυτές, στις οικονομικές και εταιρικές σχέσεις και θέλει να κρατήσει αμύωτη την ορμή για τη σύναψη οικονομικών εταιρικών σχέσεων που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, όπως προβλέπουν τα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2008. Η Προεδρία προσπάθησε να διευκολύνει την διεκπαιρέωση κάποιων εκκρεμών συμφωνιών EPA και έχουμε υπογράψει επίσημα με την από Γουινέα τον Ιούλιο μια τέτοια ενδιάμεση οικονομική εταιρική σχέση και μάλιστα ε, προωθούμε την πλήρη εφαρμογή τους από τις χώρες του Καριφόρουμ. Μάλιστα έχει βελτιωθεί το κλίμα από πέρυσι σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης χάρη σε μεγάλο βαθμό και στην προσπάθεια της Επιτρόπου Άστον που βοήθησε στην ε, ενίσχυση του διαλόγου με τις χώρες εταίρους. Τώρα για την ενίσχυση για το εμπόριο, αρρωγή για το εμπόριο, aid for trade. Αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει και πολύ πριν την Προεδρία μας. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο. Και τα θέματα αρρωγής και εμπορίου είναι αλληλένδετα και τα συμπεριλαμβάνουμε και στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επίσης θέλουμε να περάσουμε τη φάση της αναπτυξιακής βοήθειας στη φάση του ενισχυμένου εμπορίου. Υπάρχει και θέμα τεχνικής συνδρομής ή συνδρομής συναφούς με το εμπόριο, που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των εμπορικών μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα, οι χώρες ΑΚΕ θα εντοπίσουν τους αναπτυξιακούς, τους, τις αναπτυξιακές τους ανάγκες και θα τις κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα μια σύσφυξη του διαλόγου με τις ε, χώρες ΑΚΕ και μια συνδρομή της για να αυξήσουν το δυναμικό τους είναι πολύ σημαντικά γιατί το, εμπορικό, το εμπόριο είναι ένα σκέλος της αναπτυξιακής αρρώγης και μάλιστα η, το ύψος της βοήθειας αυτής θα είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2010 1 δισεκατομμύριο από τα κράτη-μέλη και 1 δισεκατομμύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα στην Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Γενέβη αυτό το θέμα το επισήμαναν ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες και δείχνουν ζωηρότερο ενδιαφέρον ε, για περισσότερο συντονισμό σε ό,τι αφορά τη βοήθεια τη συναφή με το εμπόριο. Αλλά αναφέρθηκαν και πολύ πιο συγκεκριμένοι τομείς ε, που χρειάζεται καλύτερο συντονισμός ή επιδέχονται συντονισμό. Αυτά. Μπορώ να ολοκληρώσω εδώ, να σας ευχαριστήσω και ελπίζω ότι στο σύντομο χρόνο που μου δώσετε να απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την ε, Σουηδό Υπουργό για την παρουσίασή της, για το έργο της κατά τη διάρκεια των 6-7 μηνών και ευχαριστώ και του συναδέλφους για τις ερωτήσεις που υπέβαλαν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πιόλινγκ. Sorry. Well, let's move for to the... Ας περάσουμε στο σημείο 4 της μερικής διάταξης τώρα. Συμφωνία για τα κόμματα πορεία μπανάνας μεταξύ Ευρωπαϊκής και Προμηθευτών Μπανάνας. Τέβιτο ε, Σόλβαν, David O'Sullivan, Γενικός Διευθυντής ε, της Σχετικής Γενικής Διεύθυνσης, θα πάρει το λόγο. As you know, Ξέρετε ότι το εμπόριο με την μπανάνα είναι ένα προβληματικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, πρόσφατα, οι Συντικοί υπάλληλοι συνεργάστηκαν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τους δεσμούς για την μπανάνα. Ξέρετε ότι οι πολιτικές αγωγές ε, ήταν ε, αντικείμενο μακρών διαπραγματεύσεων στην ΠΟΕ που έφεραν πρώτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλέ ε, χώρε τη Λατινική Αμερική που παράγουν μπανάνε, καθώ επίση και με τη ΣΥΠΑ. Το σημερινό καθεστώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι εισαγωγέ επιβάλλει σημαντικού δασμού στις μπανάνες που εισάγονται από χώρες που έχουν το καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους. Εκτός αυτού υπάρχουν ε, αδασμολόγητες ποσοστώσεις για εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ. Το προβλεπόμενο, η προβλεπόμενη συμφωνία είχε εξεταστεί όταν οι Υπουργοί ε, Εμπορίου συναντήθηκαν στο περασμένο Ιούλιο στην Ευή να εξαιρεθούν δηλαδή οι μπανάνες ελέγχθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε πολύ λεπτή θέση γιατί θα πρέπει να επιτύχει ισορροπία με το οξύ των συμφερόντων των λεγόμενων αποτελεσματικών εξαγωγών της Λατινικής Αμερικής και των χωρών ΑΚΕ που βασίζονται στα ε, πλεονεκτήματα που έχουν για τις εκλογέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα προσπαθείτε να υπάρχει ε, ένα νέο καθεστώς που θα βελτιώσει την οικονομική αποτελεσματικότητα και θα μειώσει τις κοινωνικές επιπτώσεις. Από την άλλη μεριά, οι χώρε τη Λατινική Αμερική θα πρέπει να διακόψουν οποιαδήποτε προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΑΕ. Από ό,τι κατάλαβαμε, οι χώρες ΑΚΕ μπορούν να δεχθούν την συμφωνία αυτή, ότι επιτεύχθη συμφωνία με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, αλλά οι ΗΠΑ Πολιτείας Αμερικής ακόμα δεν είναι έτοιμες να το δεχθούν. είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η συμφωνία για να μπορέσει να εκπληρωθεί και ο γύρος Δόχα και να υπάρχει τελική συμφωνία με τις χώρες ε, του Συμφώνου του Άντιαν και της Κεντρικής Αμερικής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε από την Κομισιόν πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συμφωνία αυτή. Καλωσορίζω λοιπόν τον ε, Γενικό Διευθυντή κ. Σάλιβαν και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πράγματι Πρόεδρε, νομίζω ότι <laughs> συνοψίζετε πάρα πολύ καλά την κατάσταση και τα θέματα που διακυβεύονται. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία στη Γενέβη για το μπανάνες. Ο πρώτος λόγος είναι αυτά τα πολλά πάνελ που χάσαμε και το γεγονό ότι ακόμα δεν ε, πληρούμε τις υποχρεώσεις μας τυπικά. Και αυτό στην ε, Γενέβη μας πλήττει και πλήττει και την αξιοπιστία μας βέβαια. Δεύτερον όμως, πρέπει να πετύχουμε συμφωνία γιατί στις διαπραγματεύσεις για την ατζέντα της ανάπτυξης υπάρχει ένας σημαντικός στόχος. Ότι δεν θέλουμε δηλαδή οι μπανάνες να θεωρηθούν τροπικό προϊόν. Αυτό που κάναμε δυο βέβαια γιατί ε, κάπως είναι τροπικό προϊόν. Το γεγονός είναι όμως ότι η τα τροπικά προϊόντα θα πληγούν σημαντικότατα. Λοιπόν, εάν οι μπανάνες το τροπικό προϊόν, θα περικοπούν οι δεσμοί πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό σχετίζεται με το θέμα ε, τότε χρειαζόμαστε βέβαια ειδική ε, αντιμετώπιση μπανάνα μπανάνας στον ΠΟΗ για να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερες πληγές και πλήγματα για το καθεστώς ιδιωτέρων προτιμήσεων των χωρών ΑΚΕ. Ο κατάλογος των τροπικών προϊόντων θα πρέπει να συμφωνιστεί στην, ε, στο γύρο αυτό που προανέφερα και εμείς έχουμε σημαντικό συμφέρον να μην συμπεριλαμβάνει ο κατάλογος αυτός προϊόντα που εμείς δεν τα θεωρούμε τροπικά προϊόντα. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον αναβόστο, για την ντομάτα, κατά πόσο αυτά είναι τοπικά προϊόντα ή όχι, αλλά πάντως στη Γενέβη θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε έναν κατάλογο. Και αυτό που θέλουμε είναι να μην συμπεριλαμβάνει αυτός ο κατάλογος προϊόντα με τα οποία θα πληγούν η παραγωγή στις χώρες ΑΚΕ. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της υπονόμευσης των προτιμήσεων. Οι χώρες και θέλουν βέβαια να έχουν περικοπές σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να ε, συμφωνηθεί. Η διαπραγματευτική ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί είναι πάρα πολύ λεπτή. Αφενός έχουμε την επίλυση των διαμαχών και το διαφωνείο την ανάγκη να έχουμε ειδική συμπεριφορά για τις μπανάνες και το άλλο είναι ο κατάλογος των τροπικών προϊόντων και ο κατάλογος των μειώσεων των προτιμήσεων. Διαπραγματευτήκαμε το τελευταίο έτος και μπορώ να πω ότι με τις χώρες Λατινικής Αμερικής και με τις χώρες ΑΚΕ πετύχαμε μια συμφωνία Όσον αφορά τις μπανάνες, πώς θα τις αντιμετωπίζουμε δηλαδή, Και στα πλαίσια του GDA αυτή η δική συμπεριφορά θα είναι τμήμα της δέσμης. Συμφωνήσαμε μεταξύ ημών και της Λατινικής Αμερικής στο κατάλογο των τροπικών προϊόντων και συμφωνήσαμε επίσης για το τα προτιμησιακά προϊόντα μεταξύ ημών των χωρών της Λατινικής Αμερικής και των χωρών ΕΚΕ. Αυτός ο γύρος ε, μπορεί τώρα να ε, μονογραφεί. Θα πρέπει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και να υπογραφεί μετά. Θα σας υποβληθεί δηλαδή μόλις φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Υπάρχουν δύο δυσκολίες που αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι ότι ο κατάλογος τροπικών προϊόντων συμπεριλαμβάνει κάποια προϊόντα που δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με άλλες χώρες του ΠΟΕ δηλαδή Αμερικής, Καναδά κλπ. Και υπάρχουν διαπραγματεύσει αυτή τη στιγμή μεταξύ των χωρών τη Λατινική Αμερική και εκείνων των χωρών. Για να μπορέσει να τελειοποιηθεί ο Εμείς θέλουμε όλα αυτά να ολοκληρωθούν το γλυγορ... ταυτόχρονα, αλλά δεν είναι αυτό τόσο απαραίτητο εφόσον σταθεροποιηθεί ο κατάλογο για τα τροπικά προϊόντα που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει με τις νομές πολιτικής Τους προσφέραμε τη δυνατότητα να συσχετιστεί με όλη αυτή τη δέσμη για τις χώρες Λατινικής Αμερικής. Εκείνοι προτίμησαν να περιμένουν, να μας δώσουν δυνατότητα να διαπραγματευτούμε με τις χώρες Λατινικής Αμερικής και μετά είπανε θα έχουν ξεχωριστή συμφωνία που τη συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Η κύρια δυσκολία που έχουμε είναι ε, η νομική διατύπωση του κειμένου. Εγώ έχω ξαναπεί εδώ, δεν είμαι δικηγόρος. Και ε, είμαι κατά βάση υπέρ της σχολής που λέει ότι δεν πρέπει να πληρώνει κανένας το δικηγόρο να του λέει τι θα κάνει. Από την άλλη μεριά προετοιμάζουμε ε, αυτό το έγγραφο μαζί με τους υπερογνώμονους ε, των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής που είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ ε, λεπτομερείς και όπου το λέμε ξεκάθαρα υπάρχει πάρα πολύ ε, δυσπιστία από όλε τι πλευρέ ο καθένα που θα ρωτήσει θα σα πει ναι, μα εμεί νομίζαμε ότι αυτό είχε ήδη λυθεί εδώ και 10 χρόνια ή το άλλο εδώ και 15 χρόνια το είχαμε τελειώσει σωστά. Υπάρχει πολλή δυσπιστία λοιπόν. Ελπίζουμε όμω θα μπορέσουμε με τη ΣΥΠΑ να πετύχουμε κάποια ε, γλώσσα κοινή τις επόμενες μέρε φαντάζομαι θα πετύχουμε τη συμφωνία αυτή αλλά ίσως είναι πολύ αργά για την παρουσίαση αυτής της δέσμης των μέτρων στο Συμβούλιο στο Γενικό Συμβούλιο για τον ΠΟΕ αυτό το θέλαμε γιατί θέλαμε αυτή η δέσμη δηλαδή η συμφωνία για την μπανάνα η συμφωνία για τον κατάλογο τροπικών προϊόντων για την μείωση των προτιμήσεων και την τελική ρήτρα που θα λέει πώς θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον οι μπανάνες θα πρέπει να σημειωθεί από όλα τα μέλη για να μην έχουμε άλλα προβλήματα στο μέλλον. Το γράψαμε στην μεσαία διάταξη του Γενικού Συμβουλίου της 17 7ης Δεκεμβρίου λυπούμε ότι θα ε, φοβούμε μάλλον ότι δεν θα προφτάσουμε να μπορέσουμε να τελειώσουμε τι διαδικασίε. Θα παραμείνει το θέμα σήμερα στη διδάξη. Θα κάνουμε μια έκθεση του πού βρισκόμαστε. Νομίζω ότι εν δυνάμει είμαστε δυνατότητα να θεωρηθούν τα κείμενα που έχουμε συμφωνήσει με του συναδέλφου από την Αμερική και για την Πανάνα και για το τοπικό πρόοδο και για την ε, μείωση των προτιμήσεων. Να τα βάλουμε δηλαδή κάπου στην άκρη και να πούμε αυτά έχουν συμφωνηθεί. Και όταν συμφωνήσουμε και τι είπα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε να περάσουμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και μετά να το φέρουμε εδώ στο Συμβούλιο εδώ και στο Κοινοβούλιο για να συμφωνηθεί. Στην αρχή είπατε ότι είναι πολύ πλοκές διαπραγματεύσει. Είναι πάρα πολύ πολύ πλοκές διαπραγματεύσει αυτές. Καμιά φορά μου το σε ο με σκάκι σε τρει διαστάσει. Αλλά τώρα πραγματικά έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ σε αυτό που θα είναι τελικά ένα... Α, ιστορικό αποτέλεσμα που οδήγησε σε τεράστια προβλήματα στο, το παρελθόν, έφερε αντιμέτωπες στις φτωχότερες χώρες, με τις φτωχότερες χώρες. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ να βρούμε τώρα αυτή τη συμφωνία και ελπίζω θα έχουμε μια ισορροπημένη λύση που θα ε, δώσει τέλος σε όλα αυτά τα προβλήματα του παρελθόν. Θα είναι σημαντικό Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ΠΟΕ και σημαντική συμβολή για το GTA, γιατί θα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις αυτές για την ανάπτυξη. Οι διαπραγματεύσεις που αυτή τη στιγμή δεν προχωρούν πολύ καλά στη Γενέβη. Όσον αφορά τη διάσταση ΑΚΕ, δεν υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμό. δεν γνωρίζουν ότι μάλλον είναι το καλύτερο που μπορούσε να επιτευχθεί. Καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει η μπανάνα να είναι τροπικό προϊόν. Έχουν κάποιο συμφέρον για τον κατάλογο που συμπεριλαμβάνει και άλλα προϊόντα που του ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και όπως είπατε και εσεί πρόεδρε, συμφωνήσαμε πάνω σε ένα πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε αυτό το VMM όπως λέγεται και ένα προπολογισμό 200 εκατομμυρίων που θα διευκολύνει τις προσαρμογές για τις ε, χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνα. Και με αυτή τη βάση οι συνάδελφοι αν και μπορούμε να δεχθούν ότι το αποτέλεσμα των προαπτήσεων ήταν οικονομικό. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Uh, about... Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε μια διεξοδική ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές μπανάνας. Θα περάσουμε σε ένα γύρο ερωτήσεων. Η κυρία Μινέμπος Κούρτ από τους σοσιαλιστές. Goedemorgen. Eh, Σας ευχαριστώ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής, αλλά είμαι πρόεδρος αντιπροσωπείας ε, για την Κεντρική Αμερική και είμαι και σοσιαλίστρια επιπλέον. Μετά την ενημέρωση που μας κάνετε, ανέκυψαν κάποια ερωτηματικά. Κάτι που επισήμανε η ίδια Προεδρία είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών. Εσείς ε, δεν το ε, αναφέρατε κύριε Σάλιβαν. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις ε, των συμφωνιών αυτών στις χώρες της αναπτυσσόμενες. Και κάτι άλλο που είπατε για τις χώρες ΑΚΕ, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Είπατε ότι οι χώρες ΑΚΕ συμφωνούν. Αλλά γιατί, τι συμφωνούν, έχουν κανένα όφελος, βελτιώνεται η κατάσταση για αυτές. Και για την Κεντρική Αμερική, το θέμα είναι πολύ σημαντικό σε διαφορά τη συμφωνία σύνδεσης με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής. Ποιε θα είναι οι συνέπειε του για τι ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσει στην περιοχή αυτή. Λυπούμε αν ε, παραπείσα το όνομά σου κυρία Μποσκούρτ. Ο Ντέβιντ Μάρτιν. <laughs> Μένω στον πειρασμό να το ρωτήσω θα επαναλάβει όλα αυτά που είπε ο Ντέιβιτ. Ήταν σαφή βέβαια όσα μας είπε και τώρα καταλαβαίνω πολύ καλύτερα το θέμα της μπανάνας γιατί από την συνεδρία τη προηγούμενη εβδομάδα με τις χώρες ΑΚΕ κατάλαβα ότι δεν ήταν και πολύ ικανοποιημένε ούτε αισιόδοξε για τη συμφωνία. Ε, εσύ τι εντύπωση αποκόμισες, Ντέιβιντ, από τις συνομιλίες με τις χώρε ΑΚΕ. Τι διαμάχες υπάρχουν και τι διαφορές Υπάρχει συνένεση μήπω για κάποιο σημείο και πού. Τώρα για το μηχανισμό αυτό το, της προσαρμογής. Έχει γίνει κάποιος, κάποια μελέτη επιπτώσεων. Ή είναι απλώ ε, ένα νούμερο που δώσαμε. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε και αν σας αρέσει. Ή μήπως έχει γίνει μια μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις, άμεσες επιπτώσεις αυτής της μείωσης των δασμών για τις χώρες ΑΚΕ. Ο Κατέρα Ρίφα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνω όλα από τη συμφωνία. Θέλω να είμαι συνετός και μετριοπαθής. Από ό,τι ξέρω, αυτό το θέμα ε, επηρεάζει και τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Η Τσικίτα κέρδισε μια υπόθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περισσότερες ε, μπανάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης από εκεί προέρχονται, κάτι που γεμίζει τα ταμεία της Τσικίτα. Οπότε μια τέτοια συμφωνία ουσιαστικά θα διευρύνει αυτή την κατάσταση. Βέβαια στο πάνελ ε, φαίνεται ότι δεν πέρασε αυτή η υπόθεση, αλλά είχα την αίσθηση ότι δεν έγινε καμία προετοιμασία ούτε συμφωνία του Κοτονού ούτε στο Λομέ προηγουμένω. Είπαμε στους μπανανοπαραγούς να προετοιμαστούν γιατί το μέλλον θα ήταν περίπλοκο και δύσκολο. Τώρα προτείνεται διαφοροποίηση για τους μικροπαραγωγούς, αλλά πώς θα υλοποιήσουν αυτή την διαφοροποίηση, γιατί ήταν απροετοίμαστοι. Στο μηχανισμό προσαρμογής, το BAM, δόθηκαν 110 εκατομμύρια καταρχήν, μετά 104 ή 194. Δεν ξέρω αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω. Σήμερα τι γίνεται, τι γίνεται με αυτά τα συνοδευτικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πέραν των συνοδευτικών μέτρων που είναι συγκυριακά και προσωρινά. Υπάρχει πολιτική, οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν για να βοηθηθούν αυτοί αυτές οι χώρες και η μπανανοπαραγωγή για να μην μειωθεί η ανάπτυξή τους και να μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό των μεγαλοπαραγωγών από τη ζώνη ΟΛΑ. Thank you. Also from Merci, Monsieur le Président. συνεχίζω τις προηγούμενες παρατηρήσεις του Καντέρα Ριφ. Μας παρουσιάσετε την πτυχή υπό το πρίσμα των διπλωματικών διαπραγματεύσεων και της νομικής διάστασης. Αλλά δεν μιλήσατε και πολλά για τα οικονομικά. Βέβαια αυτό το στόχο έχει το ΜΠΑΜ, αυτός ο μηχανισμός προσαρμογής. Οι δασμοί θα περιοριστούν κατά 35% για τις χώρες ΑΚΕ και υπάρχει κίνδυνος μείωση μέχρι 80% αν οι μπανάνες μπουν στην κατηγορία των τροπικών προϊόντων. Ποια θα είναι η συνέπεια όμως για την ευρωπαϊκή αγορά και πώς θα επηρεάσουν τις εξαγωγές των χωρών ΑΚΕ. Γιατί έγινε μια μελέτη, όπως είπε ο Ντέιβιτ Μάρτιν, με αυτό το αντικείμενο. Το ΜΠΑΜ, αυτός ο μηχανισμός προσαρμογής, υποτίθεται θα αντισταθμίσει κάποιες απώλειες, αλλά αναφέρθηκε ένα είδος ε, ανακύκλωση μετατροπής σε τι καλλιέργεια θα μπορούσαν να στραφούν οι μπανανοκαλλιεργητές αν είναι να αλλάξουν. Αλλά υπάρχουν τεράστιοι οικονομικοί κραδοσμοί για τους ε, παραγωγούς ΑΚΕΣ ό,τι αφορά το κύκλο εργασιών τους. Και θα υπάρξει αντίκτυπος και στις ε, υπεραπόμακρες περιοχές, στους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς. Και τι μέλη γενέστε. David Μάρτιν, σύντομο συμπληρωματικό σχόλιο. Δεν ξέρω, γιατί όταν είπε για την Τζικίτο Ακαντήρ, ε, θυμήθηκα και την ερώτηση αν ο Παναμάς έχει προσυπογράψει αυτή τη συμφωνία που ξέχασα πριν. Γκουε. Μία μικρή ερώτηση από αυτό. Η συμφωνία για την μπανάνα σχετίζεται ίσως με τον κατάλογο για τα τροπικά προϊόντα, αλλά ίσως και κατά πόσον οι χώρες εκεί αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται και άλλα τροπικά προϊόντα να συμπεριληφθούν στο κατάλογο αυτό, να εξετάσουν δηλαδή θα γίνει, να μειωθούν οι δασμοί κλπ. Η σύναψη της συμφωνίας αυτές ε, έχει λοιπόν μεγάλη συμφωνία και για άλλα εμπορικά προϊόντα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα τροπικά. Okay, thank you. Okay. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον Ντέβιντο Σάλιβεν για να απαντήσει. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της συμφωνίας αυτής. Σίγουρα επιτείνεται η διάβρωση των προτιμήσεων που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι χώρες ΑΚΕ. Και πολύ φοβούμε ότι μια τέτοια διάβρωση είναι αναπόφευκτη για τις προτιμήσεις. Και αν χρειαστεί να συμφωνήσουμε με τους ε, Λατινοαμερικάνους προμηθευτές μπανάνας και υπάρχουν και βιομηχανικά συμφέροντα που δεν θα πρέπει να τα ξεχνούμε, αλλά μιλούμε για φτωχέ χώρε που εξαρτώνται από τι εξαγωγέ αυτέ και οι εξαγωγέ αυτέ εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ευημερία των λαών του. Και έχω μια αντιπαράθεση εδώ μεταξύ των φτωχών Λατινοαμερικάνων κατά των φτωχών ε, των χωρών ΑΚΕ. Ακόμη όμως και με το δασμό 176 που ισχύει τώρα, οι χώρες ΑΚΕ, η μπανανοπαραγωγή των χωρών ΑΚΕ διατήρησαν και μερικές φορές ε, ε, ανέβασαν το μερίδιό τους. Βέβαια, αν είχαμε υψηλότερους δασμούς ε, από το 176 θα είχαμε... Βέβαια, πριν μάλλον να φτάσουμε στο 176, οι προβλέψεις αν θα το εφαρμόζαμε ήταν πολύ ζωφερές, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι απεσιόδοξες προβλέψεις με το 176. Βέβαια, υπάρχουν πολλέ δυνατότητες που προβλέπονται στο μηχανισμό προσαρμογής για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ε, δυνατότητα των παραγωγών να εξυγχρονίσουν ε, και να βελτιώσουν την παραγωγή τους στις χώρες ΑΚΕ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς για τις χώρες ΑΚΕ. Βέβαια, το μέλλον είναι απρόβλεπτο. Τουλάχιστον δεν μπορούμε με ακρίβεια να προβλέψουμε το ποσό. Πάντως οι χώρες ΑΚΕ απρόθυμα μεν, αλλά δέχτηκαν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουν κάποια εχέγγυα για το μέλλον. Κάποια εχέγγυα για ελεγχόμενη και αποδεκτή μείωση ε, των δασμών που δεν θα γίνει φυσικά εν μία νυχτή αλλά θα γίνει σε μία περίοδο 6-7 ετών. Και επίσης θα δοθούν κάποια εγγύηση ότι αφορά την ε, διάβρωση των προτιμήσεων, όπως ανέφερε και ο κύριος Σούλτς. Δυστυχώς διαφωνώ με τον κύριο Άριφ. Δεν συμφωνώ ότι δεν προετοιμάσαμε τους ε, ομολόγους μας από τις χώρες ΑΚΕ για αυτό το δεχόμενο. Και περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ δόθηκαν ε, ως αρρωγή στους μπανανοπαραγωγούς στις χώρες ΑΚΕ με από το Αναπτυξιακό Ταμείο και τα 200 εκατομμύρια ευρώ είναι επιπλέον των 800 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη δόθηκαν στους μπαναναπαραγωγούς για να αντιμετωπίσουν τους κραδασμούς και να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Και μάλιστα το Αναπτυξιακό Ταμείο βοήθησε τις χώρες ΑΚΕ για να κάνουν όλες αυτές τις προσαρμογές και να ε, προετοιμαστούν στη νέα κατάσταση που ήταν ε, αναπόφευκτη στα πλαίσια και των διαπραγματεύσεων για την DDA. Και μάλιστα στο 10ο Αναπτυξιακό Ταμείο έχουμε 23 δις ε, που θα προσφερθούν ως ε, ενίσχυση στις χώρες ε, και για να στηρίξουν την οικονομική τους ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση. Υπάρχουν αυτά τα κονδύλια και θα δοθούν για τις χώρες αυτές. Οπότε είναι σχετικό το νούμερο των 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι συμπληρωματικό ποσό στο υπάρχον κονδύλιο του Αναπτυξιακού Ταμείου που είναι πολύ μεγαλύτερο και θα βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να αντιμετωπίσουν ε, το κόστος ε, προσαρμογής στην εγκατάσταση και διαφοροποίησης. Για τους Ευρωπαίους παραγωγούς οι Ευρωπαίοι μπανανοπαραγωγοί είναι αυτοί που λαμβάνουν τις περισσότερες επιδοτήσεις. Έχουν ε, τους υψηλότερους συντελεστές επιδότησης από τους άλλους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων σε καμία περίπτωση δεν τους παραμελήσαμε. Υπάρχουν προγράμματα για τους Ευρωπαίους μπανανοπαραγωγούς. Μην ξεχνούμε όμως ότι οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών από τη Λατινική Αμερική και αυτοί προέρχονται από αναπτυσσόμενες και φτωχές χώρες. Και μάλιστα οι χώρες αυτές ε, θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή που έχει κρατήσει τόσα χρόνια με υψηλότατους δασμούς, με πολλές προτιμήσεις εις βάρος τους ή πολλές αρρωγές τους έχουν φέρει σε δυσμενή κατάσταση και εξού και η διαμάχη στη Γενέβη και αυτή η διαφορά που προσπαθούμε τώρα να διευθετήσουμε. Ως προς τώρα συμφωνούν λοιπόν οι χώρες ΑΚΕ. Είχαμε πραγματικά εξαντλητικές συζητήσεις. Δεν θέλω καν να υπολογίσω πόσες ώρες περάσαμε στις διαπραγματεύσεις Πόσε ανθρωπόρε ξοδέψαμε στι διαπραγματεύσει. Είχαμε ανθρώπου που του κλειδώναμε σε αίθουσε μερόνυχτα ολόκληρα. Πρώτα με ε, τους καταλόγους και τις προτιμήσεις ε, των Λατινοαμερικάνων, μετά με τις προτιμήσεις των χωρών ΑΚΕ. Προσπαθήσαμε να τους αναμίξουμε σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Και δεν σας λέω ότι όλοι θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και δεν θα βρεθεί κάποιο παραγωγό τη χώρα ΑΚΕ που θα έχει δυσαρεστηθεί. Πάντω σα υπόσχω, σα δίνω το λόγο μου, του αναμίξαμε σε όλες τις φάσεις διαπραγμάτευση. και εγώ πιστεύω ότι απρόθυμα μένα, αλλά παρόλα αυτά συμφώνησαν με την πρόταση αυτή, γιατί αναγνώρισα ότι είναι ο μόνος τρόπος για να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση και να ικανοποιηθούν κάπως ό,τι αφορά τη διάβρωση των ποσοστώσεων των προτιμήσεων συγγνώμη, και να βρεθεί μια λύση για τις μπανάνες στο DDA. Με τους Λατινοαμερικάνους Υπάρχει ήδη υπογραφή με όλους τους παρανοπρομηθευτές ε, που απολαμβάνουν το καθεστώς του πλέον ευνομένου κράτους. Βέβαια δεν είναι οργανωμένοι, προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα, οι πιέσεις είναι διαφορετικές, αλλά και πάλι χάρη στις ε, καταπώνητες προσπάθειες ε, του διαπραγματευτή μας στη Γενέβη καταφέραμε να προσυντεριστούμε όλους μας τους εμπορικούς εταίρους και έχουμε ένα κείμενο με συμφωνημένο κατάλογο προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συνέπειες ε, για τις ε, συμφωνίες ε, της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου, αν συμφωνήσουμε για τις μπανάνες πολυμερό στη Γενέβη, λύνονται τα χέρια μας για να ολοκληρώσουμε και τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία και το Περού. Γιατί εκεί και πάλι οι μπανάνες είναι το πιο νευραλγικό σημείο. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε την καλύτερη μας προσφορά για τις μπανάνες. Γι' αυτό και έκαναν πίσω οι εταίροι μας, περιμένοντας μια καλύτερη προσφορά. Και από αυτή την άποψη, μια θετική παρενέργεια μια τέτοια συμφωνία για τις μπανάνες θα είναι να απεμπλέξει τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τι χώρε Κεντρικής Αμερικής και με το Περού και την Κολομβία. Κύριε Σούλτς, κύριε Σόλτς, δεν ξέρω αν κατάλαβα την ερώτησή σας για τα τροπικά προϊόντα. Ρωτήσατε αν θα έχουμε πρόβλημα με άλλα προϊόντα που θα ενταχθούν στον κατάλογο των τροπικών. Πάντως, ένας από τους στόχους των διαπραγματεύσεων είναι να σταθεροποιήσουμε, να συμφωνήσουμε και να κλειδώσουμε, θέλετε, ε, να οριστικοποιήσουμε τον κατάλογο των τροπικών προϊόντων μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις. Γιατί κάποιοι προμηθευτές ΜΕΚ αυτών των προϊόντων είχαν μια πολύ γενική εικόνα για το τι εστί τροπικό προϊόν και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς Ευρωπαίους παραγωγούς που για μας δεν είναι τροπικά του παράγοντα εύκρατε ζώνε. Λοιπόν, προσδιορίσαμε τον κατάλογο, τον οριστικοποίησαμε, μπορούμε να τον δεχτούμε και εμεί και οι Λατινοαμερικάνοι. Οπότε, κατά κανόνα, έχει αποκρισταλωθεί ω τμήμα των γεωργικών συμφωνιών στο πρόγραμμα αναπτυξιακών στόχων και συμφωνιών της στόχας αποτελέσει τμήμα αναπόσπαστο και κεκτημένο των γεωργικών διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το ε, επιδιώξαμε πάση θυσία. Αντιλαμβάνομαι και το σχόλιο για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και μάλιστα και από το πρίσμα των χωρών και μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε και μακάρι να μην το κάνατε θα μας έλεγαν οι χώρες ΑΚΕ αλλά μας δεσμεύουν νομικά τα πάνελ. Οπότε θέλουμε και οι Λατινοαμερικάνοι να προσυπογράψουν το DDA για τις μπανάνες. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε διαπραγματεύσει και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Επίσης έχουμε και ηθικό καθήκον απέναντι στις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής που εδώ και πολύ καιρό αισθάνονταν πολύ δυσμενή μεταχείριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πια θα ξεπεραστεί. Θα καταλήξουμε σε δίκαιο και ισορροπημένο αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους και τις χώρες Λατινικής Αμερικής και τις χώρες ΑΚΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαπραγματευτικό σώμα αλλά και τους Ευρωπαίους μπανανοπαραγωγούς που έχουν φυσικά συμφέροντα που θέλουν να διαφυλάξουν. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια που μας δώσατε. Και ευχαριστούμε επίσης για το γραπτό κείμενο που μας ε, ε, υποβάλλεται γιατί μας δίνει πραγματικά πολύ σαφείς ιδέες για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι προοπτικές τους. Περνάμε στο σημείο 5. Επιπτώσει παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στι αναπτυσσόμενε χώρε και στην αναπτυσσιακή συνεργασία. Ανταλλαγή απόψεων προβλέπεται για αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε η Επιτροπή Ανάπτυξης αποφάσισε να προετοιμάσει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το εν λόγω θέμα και η δική μας Επιτροπή αποφάσισε να γνωμοδοτήσει. Από τότε που πέρασε η χρηματοπιστωτική κρίση από τη ΣΥΠΑ σε εμάς, πέρσι το Σεπτέμβριο, οι επιπτώσεις της κρίσης αυτές γίνονται όσο πάει και πιο αισθητέ και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εμπόριο, άμεσες εξωτερικές επενδύσεις. Υπάρχουν ε, τώρα κάποιες ενδείξεις για ανάκαμψη, αλλά οι πιο φτωχές χώρες εξακολουθούν να υποφέρουν από την παγκόσμια ύφεση. Γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε τη γνωμοδότηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρία Μουνή. που είναι η συντάκτα τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή μα και που θα μα εισαγάγει το θέμα. Μαρία, έχετε το λόγο. Eh, señor presidente. Efectivamente, como usted dice, la economía global está dando signos. Η παγκόσμια οικονομία δίνει μηνύματα ανάπτυξης, αλλά οι αναπτυσσόμενες χώρε αντιμετωπίζουν σοβαρέ επιπτώσεις περιπτώσεις ε, που απειλούν και τις κατακτήσεις των τελευταίων ετών. Κυρίως ε, όλη την πρόοδο που, έχουν γίνει, που έχει γίνει για την καταπολέμηση της στόχιας και την προσέγγιση των στόχων της χιλιετίας. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές όχι μόνο αποτελούν το επίκοντρο της κρίσης, αλλά μειώνουν και τις δυνατότητες συναλλαγής των αναπτυσσομένων χωρών. ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών με τη συνένεση της Ουάσιγκτον μειώνεται η ζήτηση και σε σχέση με το 2007 η ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών μειώθηκε κατά ένα τέταρτο και κατά ένα τρίτο σε σχέση με το 2007. Σύμφωνα με την ΔΟΕ, 200 εκατομμύρια άτομα θα προσθεθούν στο 1 δισεκατομμύριο 300.000 άτομα που εργάζονται με κάτω από 20 ε, δολάρια το μήνα. η μείωση των τιμών του πετρελαίου κατά 20% μείωσε τα ισοζύγια των αναπτυσσομένων χωρών και στο ισοζύγιο εξαγωγών θα έχουμε μέχρι και 17% αρνητικό ισοζύγιο για τις εξαγωγές από τις αφρικανικές χώρες. Αυτό θα έχει επιπτώσεις και στον δανεισμό και στη χρέωση. Η στάση των άλλων χωρών γίνεται προστατευτική και θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές τις αγορές ε, για να παλέψουμε κατά της ύφεσης ε, και να εξωθήσουμε την ανάπτυξη τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι, ροές, οι δημοσιονομικές ροές προς τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περιοραστεί και το FMI e, μόνο το 1 τρίτο των ε, αναγκών χρηματοδότηση αυτών των χωρών θα καλύψει. Το εξωτερικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 2% του ΕΠ τα τελευταία χρόνια και τα έσοδα από τις απτεβάσματα των μεταναστών θα μειωθούν κατά 7%. Ξέρουμε ότι αυτού του είδους τα, τα εισαγόμενα κεφάλαια καλύπτεται το 6% του ΑΕΠ αυτών των χωρών. Η έκθεση του κυρίου Γκερέρο στην Επιτροπή Ανάπτυξης είναι πολύ ολοκληρωμένη και πλήρης. Ε, θα έπρεπε όμως ε, σε αυτήν την ε, γνωμοδότηση σε αυτήν την έκθεση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γνωμοδότηση που εγώ έχω υποβάλει στις εξής, στις γραμμές συνοχή των πολιτικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε η εμπορική απολευθέρωση να γίνεται στο βαθμό που συμβάλλει στην ανάπτυξη και η οποία θα είναι ουσιαστική όσο τη θέλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να ενσωματωθούν και κοινωνικές πτυχές όπως ε, οι αξιοπρεπείς εργασίες. Θα πρέπει να έχουμε επίσης ε, πολυμερότητα απαιτώντα την ολοκλήρωση του γύρου της ε, ΔΟΑ και επίσης τη σύναψη συμφωνιών σαν αυτή για την μπανάνα. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αξιοπρεπή απασχόληση, μείωση των τιμών κατανάλωσης και ένα δισεκτήριο εκατομμύριο της ε, ε, Κομισιόν και των κρατών μελών όπως έχει ήδη συμφωνηθεί θα πρέπει να <coughs> δοθούν ως χρηματοδότηση για την ενίσχυση του εμπορίου αυτών των χωρών και τη μείωση της στόχιας. Και θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται σχετικά με τον προορισμό αυτών των κονδυλίων. Η Κομισιόν θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο δυναμικό και φιλόδοξο στα διεθνή όργανα να λάβει υπόψη ε, και τα απορίσματα της Επιτροπής ε, Στήλιτς για τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες θα πρέπει να ζητήσουμε την ανάπτυξη τοπικών τραπεζών αναπτύξεως. Ενίσχυση επίσης των συναλλαγών νότου-νότου. διότι οι διμερείς ε, συμφωνίες δεν δίνουν σήμερα αυτά αποτελέσματα, γι' αυτό θα πρέπει να υποστήριξουμε εναλλακτικέ λύσεις. Πιστεύω ότι με αυτές τις παρατηρήσεις θα ενισχύσουμε την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης που ήδη είναι αρκετά πλήρης. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ερώτηση για τις λιγότερο από Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας Αλεξάρ Τζόνς. Over there on my right, please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Um, on behalf... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξονόμη το Επιτροπής. Ήθελα να σας πω ότι χαιρετίζουμε αυτή την έκθεση που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή σήμερα το πρωί βέβαια και την γνωμοδότηση που μόλις παρουσιάστηκε σε εμάς. Η Κομισιόν συμφωνεί με πολλές από τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες που παρουσιάζεται στην έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν ε, αναγνώρισε γλίγορα ότι η κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες Ξέρετε ότι υπέβαλε μία ανακοίνωση μετά την ε, διασκορσή του G20 στο Λονδίνο με μία σειρά μέτρων για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση. Τα μέτρα αυτά υποστηρίχθηκαν σε μεγάλο ποσοστό από το Συμβούλιο φέτος το Μάιο και ορισμένα τα κύρια μέτρα αφορούν τις ε, ε, δεσμεύσεις uh, του ODA και ότι υπάρχει ένα μέσο που αναφέρεται στο λεγόμενο μέσο για vulnerability flex για να δώσει χρήματα ε, και δημοσιονομική ενίσχυση στις χώρες που έχουν προβλήματα. Και πολλές από τις χώρες αυτές θα βοηθηθούν από την ε, γλίγορη αυτή βοήθεια μέχρι το τέλη του έτους. Φέτος και άλλες μέχρι το 2010. Ε, επίσης θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τους άλλους χώρες τη φοροδιαφυγή, τους φορολογικούς παραδείσους και να δώσουμε συμπληρωματικούς πόρους για το λεγόμενο ε, ταμείο για ενίσχυση για τις υποδομές. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που ίσως έχουν περισσότερα ε, πληροφορίες για το θέμα των ε, εμπορικών σχέσεων. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος, να ακούσω και τα άλλα μέλη της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής. Who is willing to take the floor? I'm sorry, Chairman, but, uh... Λυπούμε, αλλά δεν έχουμε κανέναν να τη διεύθυνση του εμπορίου. Γιατί αυτή είναι η έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Uh, okay. Uh, so I'll now, I now give the floor to other... Καλά, να δώσω το λόγο τότε στα μέλη της Επιτροπής μας. Θέλει κανείς να σχολιάσει. May I call your attention, please? David Martin. Μα David Martin. I think, uh, first I would like to... Θα ήθελα κυρίως να συγχαρώ τη Μαρία για την uh, πολύ εύστοχη έκθεσή της. Η ανάλυση της uh, ήταν οξυδερκέστατη και σαφέστατη. Τι να πω, τι να προσθέσω. Και μετά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλό θα ήταν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα εμπορίου περισσότερο, στην πτυχή του εμπορίου, παρά να μιλούμε για τα θέματα που είναι αρμοδιότητα της, ανά... της Επιτροπής Ανάπτυξης καλό θα ήταν να αφήσουμε ανοιχτέ τι αγορέ μα ε, στα εμπορικά προϊόντα αυτών των αναπτυσσομένων χωρών και να προωθήσουμε το εμπόριο με τι χώρε αυτέ. Να εξετάσουμε και τα φυτογειονομικά μα μέτρα. Σε καμία περίπτωση βέβαια να μην υπονομεύσουμε τη δημόσια υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ελαφρύνουμε κάπως τεχνικές προδιαγραφές, διευκολύνοντας την πρόσβαση αυτών των χωρών στις αγορές μας. Μα ενδιαφέρει και η συνέπεια και η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών μα Κρίμα που το εμπόριο δεν περιλαμβάνεται ω αναπόσπαστο στο τμήμα τη αναπτυξιακή μα πολιτική. Γιατί είναι αλληλένδετο το εμπόριο με την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να μα λέει η Γενική Διεύθυνση του Εμπορίου αυτό είναι θέμα ανάπτυξη, εμεί δεν έχουμε καμία σχέση. Θέλουμε συντονισμό, συνεργασία και συνάφεια μεταξύ των προσπαθειών των δύο Γενικών Διευθύνσεων. Πολύ σωστά, Ντέιβιτ. Σίγουρα το εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί ρηκτό τμήμα της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Μαρία, θέλεις να προσθέσεις κάτι για να ολοκληρώσουμε. Όχι, ευχαριστώ. Και για τα σχόλια της Κομισιόν και για τον Τζέβιν Μάρτιν. Θα ετοιμάσω ένα πρόχειρο για το οποίο να συζητήσουμε και μετά να έχουμε και τις τροπολογίες ε, τη Επιτροπής, ελπίζω όχι πολλές, λόγω της συνένεση που προσεγγίσαμε τώρα, δεν φαντάζομαι μετά υπάρξουν διαφωνίε. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα για την εξέταση της έκθεση υπάρχει στον φάκελό σας. Η πρώτη συζήτηση έγινε σήμερα, 27 Ιανουαρίου, εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης, προθεσμία για την αποβολή τροπολογιών 2 Μαρτίου, και η αθέτηση της γνωμοδότησης. στις 23 του μηνός. And Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 6. Συνοχή της ανεψυχής πολιτικής και επίσημη αναισθητική βοήθεια συν. ΕΒΑ συν. Ανταλλαγή απόψεων. Ξέρετε ότι αυτό εισήχθη στην συνθήκη του Μαστρίχια πρώτη φορά, η συνεπιά και η συνοχή όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και νομική βάση νέα συνθήκη της Σαββόνας. Οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θα πρέπει να είναι αντιφατικές και θα πρέπει όλες να είναι επίσης ώρες. Το Σεπτέμβριο φέτος ε, η ε, Κομισιόν δημοσίευσε μια γνωμοδότηση για την σφαιρική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται στις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της συνοχής πολιτικής για την ανάπτυξη. Η πολιτική ανάπτυξη αποφάσισε να προετοιμάσει μια έκθεση ίδια πολιτικής για τη συνοχή της ανάπτυξης πολιτικής βασιζόμενη στην ανακοίνωση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική μα Επιτροπή αποφάσισε επίση να γνωμοδοτήσει. Ε, θα πρέπει να το περάσουμε πολύ γρήγορα γιατί κανονικά η συνεδρία των συντονιστών θα πρέπει να έχει αργήσει 11.30 ήδη και έχει περάσει η ώρα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Του τον εκθένω θα ήθελα να δώσω το λόγο στον τροχιά που είναι ο, ο συντάξει γνωμοδότηση για την Επιτροπή μα και θα μα συζητάει το μέλλον. Πού είσαστε παρακαλώ. Α, ναι, σα είδα. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός γιατί πέρασε η ώρα. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Μα ζήτησαν γνωμοδότηση για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, σε σχέση με το εμπόριο, γιατί αυτό που συμβαίνει σε ένα ιδιαίτερα εύρωστο οικονομικό μπλοκ του κόσμου έχει τραγικές συνέπειες σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είδαμε πρόσφατα από την κρίση του διεθνούς καπιταλισμού που έπληξε τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις φτωχές και τις ε, φτωχότερες των φτωχών. Και η κερδοσκοπή των τελευταίων δέκα χρόνων ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης ε, προκάλεσαν ολέθριες συνέπειες για τις μάζες των φτωχών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πιστεύω ότι θα πρέπει στον τομέα του εμπορίου να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια η θέση της για την αναπτυξιακή συνεργασία. Στις συνθήκες, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρανώνει την προσήλωσή της στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών και ιδιαίτερα των πιο μειονεκτικών από αυτές λέει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας ε, στις χώρες αυτές είναι προτεραιότητα της και το άρθρο 178 προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει υπόψη του στόχου του 177 στις πολιτικές της που ενδεχομένω έχουν επίπτωση σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό ήταν πριν τη δήλωση του 2005 του Προέδρου της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν ε, συνυπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Εκεί αναφέρθηκε ο στόχος της ε, καταπολέμησης της φτώχειας, ε, του υποδιπλασιασμού της μέχρι το 2015 και της εξισορρόπησης μεταξύ των δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και την προάσπιση των, του εθνικού πλούτου από τη μια πλευρά και της ανάπτυξης α, ε, της οικονομικής και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης από την άλλη. Αν κοιτάξουμε το στρατηγικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2006 και το στόχο της για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τις συμφωνίες εταιρική σχέσης, διαπιστώνουμε ότι περιορίζεται στους, ε, στην εξασφάλιση πρόσβασης για τις πρώτες ύλες και για κάποια α, προϊόντα και ζητά ισχυρού κανόνε για το άνοιγμα των αγορών, την πνευματική διοκτησία, τι υπηρεσίε, τι επενδύσει, τι δημόσιε προμήθειε και τον ανταγωνισμό. Η υπηρεσία ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίε είναι ακρογωνίω λίθο ε, τη παγκόσμια οικονομία και η απελευθέρωση αυτών των τομέων ε, θα βοηθήσει του εταίρου μα εκεί που υπάρχει χαμηλή πρόσβαση στην αγορά. Υπάρχει όμω ασυνέπεια μεταξύ των ε, στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προϋποθέσεων και των όρων που βάζει στις αναπτυσσόμενες χώρες με αυτά τα υψηπετή που περιλαμβάνει στις ιδρυτικές της συνθήκες. Υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια δηλαδή μεταξύ των δηλώσεων και των παράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα εμπορικών συμφωνιών και την πραγματική πλευρά του εμπορίου ε, αυτού με τις χώρες τα τελευταία δέκα χρόνια. θα μπορούσαμε να εξετάσουμε διάφορες πτυχές του εμπορίου. Για παράδειγμα, τη σχέση με την, την κοινότητα των άδεων και τις προσπάθειες για τις συμφωνίες εκεί. Και πρόσφατα ε, τη συμφωνία με το Καριφόρουμ. Γιατί και στη συμφωνία αυτή διαπιστώνεται μεγάλη ασυνέπεια σε εμπορικά ζητήματα μεταξύ των ε, λόγων και των προθέσεων και των πράξεων. Φαντάζομαι θα μας πει τη γνώμη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν πάντως συντάσσει τις προτάσεις της για την πολιτική και τη συνοχή της, φαίνεται ότι εσκεμμένα προσπαθεί να ε, εξοβελήσει το εμπόριο. Εμείς θέλουμε το εμπόριο να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα αυτών των, αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής και όχι συστηματικά να αποκλείεται. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, για την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ΣΥΝ λέει ότι η χρήση ε, διαφόρων διάβλων πέραν της δημόσιας ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Τι εννοεί, τι εννοεί ακριβώς σημαίνει ότι θα αναθέσει την αναπτυξιακή βοήθεια σε ιδιωτικούς φορείς, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πάντως, οι λαοί των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν πολύ κακή πείρα με τις ε, ευρωπαϊκές πολυεθνικές, για παράδειγμα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Εξαιτίας των δεινών ε, όρων που τους υποβάλλουν και την απομίζηση που υφίστανται των πρώτων υλών τους. Αυτές είναι κάποιες ε, εισαγωγικές σκέψεις για τη γνωμοδότησή μου, κύριε Πρόεδρε. Και σας λέω ειλικρινά ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αρρωγή προσφέρει σε αυτές και μεταξύ αυτής της τάσης και της ε, έμπρακτης εφαρμογής εμπορικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε μαζί μας τις ιδέες που θα προσθέσετε στην γνωμοδότησή σας. Τώρα υπάρχουν παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις από τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας. No. Δεν φαίνεται. Α, ναι, ο David Μάρτιν. Πάρα πολύ σύντομα. Γιατί τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ σωστά πρέπει να είμαστε συνεπείς στην μα πολιτική και θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε και η ε, Σουηδός υπουργό για το θέμα της πρόσβασης στα φαρμακευτικά προϊόντα γιατί καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες στην αναψυχημένη μα πολιτική για να καταπολεμήσουμε το AIDS, την ελληνοσία, φυματίωση ε, κλπ. Και καμιά φορά βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να είναι ένα θέμα που θα είναι το πιο κύριο στο νου μας. Και παρόλο που στις αντίθετες δηλώσεις ε, φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ημών και τρίτων χωρών ε, επιβάλλουμε καμιά φορά πάρα πολύ σκληρές ε, προϋποθέσεις και πολύ σκληρούς όρους που μου φαίνεται απαράδεκτο. Γενικότερα, μια από τις ιδέες που θα πρέπει να βελτιωθεί είναι το θέμα της αξιολόγησης των ε, οικονομικών επιπτώσεων. Εμένα μου φαίνεται ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο ε, δεν είναι καθόλου διαφανές, ε, δεν ξέρουν όλοι τι γίνονται η κοινότητα των πολιτών στι εν λόγω χώρες επίσης δεν ξέρει ακριβώ τι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο γενικά το θέμα τη κοινωνία των ε, πολιτών όταν μιλάμε για προγράμματα για αναπτυσσόμενες χώρε, Εγκρίνουμε πολλά, αλλά νομίζω ότι δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με του πολίτε εκεί τόπου για να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε που έχουν και ποιε είναι οι πολιτικέ που θα μπορούσαν να του βοηθήσουν γιατί καμιά φορά λέγεται ότι μεταξύ τη πραγματική πολιτική και της ε, δηλουμένης πολιτική υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί εκεί. Γενικά χαιρετίζω το γεγονό ότι υπάρχει τώρα πια μια νομική βάση για το θέμα και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση νομίζω. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι βέβαια η πρώτη παρουσίαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω κατά πόσον η Κομισιόν θέλει να κάνει κάποια σύνομη πρώτη παρατήρηση για το θέμα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι γερετίζουμε τη συζήτηση αυτή. Είναι περίεργο, αλλά ακριβώ πριν από ένα μήνα Είχαμε την ίδια συζήτηση στην Επιτροπή Ανάπτυξη και χαιρόμαστε που και άλλε επιτροπέ εκτό από την ανάπτυξη πολιτική εξετάζουν το θέμα αυτό. Θα έπρεπε να εξεταστεί από πολλέ επιτροπέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί πραγματικά το θέμα τη συνοχή για την ανάπτυξη και βοήθεια είναι και για την ανάπτυξη γενικά είναι θέμα τη Κομισιόν, αλλά είναι και θέμα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Εμεί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε παρά μόνο όταν συνεργάζονται όλα τα θεσμικά όργανα. Είναι μια υποχρέωση από τη συνθήκη η συνοχή αυτή στην ανάπτυξη. Λέχθη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μας όλες τις πολιτικές που μπορούν να έχουν επιπτώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες Το γενικό πλαίσιο ορίστηκε το 2005 όταν η Κομισιόν ανέλαβε δεσμεύσει σε 12 τομεί μεταξύ των οποίων ήταν και το εμπόριο. Το Σεπτέμβριο φέτος το η Κομισιόν εξέδωσε δύο έγγραφα για την επίσημη ενεψυχική βοήθεια. Το ένα λέγεται εδώ βλέπετε είναι η έκθεση για την ε, ε ΕΒΑ. Είναι μια πλήρης ε, έκθεση που αναφέρεται στην ε, ε πρόοδο που έχει τριφθεί στους 12 κύριους τομείς. Ίσως σας ενδιαφέρει ότι το ε, κεφάλαιο για το εμπόριο είναι το πιο μακροσκελές κεφάλαιο της έκθεσης. Ταυτόχρονα όμως ε, δώσαμε μία ε, ανακοίνωση για τη συνοχή της αναψυχής πολιτικής με στόχο να αναζωογονήσουμε την προσέγγιση μας και να είμαστε πιο ενεργοί και δραστήριοι στην προσέγγιση της συνοχής αναψυχικής πολιτικής και να αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στα θέματα της ε, ανάπτυξης όταν εξετάζουμε διάφορα θέματα της ε, κοινωνικής πολιτικής. Αυτή η έκθεση τώρα έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο και εμείς θα βασιστούμε στο μέλλον σε πέντε τομείς, δηλαδή χρηματοδότηση και ε, εμπόριο, κλιματικές αλλαγές, ε, ασφάλεια στον τομέα των τροφίμων, ε, ειρήνη και ασφάλεια. Αυτοί οι τομείς εξελέγησαν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα να καθιστούν θα τους καταστήσουμε πιο φιλικούς για την ανάπτυξη. Είναι ε, σημαντικό να σας πω ότι στην αρχή δεν υπήρχε το εμπόριο σαν μία από αυτές τις πρωτοβουλίες γιατί θεωρείται ότι έχει ήδη λεχθεί αυτό και ήδη έχουν αληφθεί δράσεις και δεν χρειάζεται να επιλεχθεί εκ νέου σαν μία από τις προτεραιότητες. Και μετά συζητήσουμε το Συμβούλιο διαφάνει ότι αυτό θα απόδιδε ένα εσφαλμένο πολιτικό μήνυμα και τώρα γι' αυτό έχει συμπεριληφθεί και θα το εξετάσουμε. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η εστίαση σε αυτούς τους ε, πέντε τομείς δεν σημαίνει ότι μειώνουμε τον αριθμό των τομείων πολιτικής που θα μας απασχολήσουν. Παραδείγματος χάρη την ε, παγκόσμια πρόκληση για την ασφάλεια τροφίμων. Αυτό δεν είναι μόνο γεωργία, αλλά και η εμπορική πολιτική, παραδείγματο χάρη, που συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτο, διακόπτε, σα παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, ναι, και, ναι, ναι, τρικλίνω. Και μέσα στα πλαίσια τη ε, ε, παγκόσμια ε, ασφάλεια για θα εξετάσει το θέμα τη αλληλείας, κλιματικές αλλαγές. Αν έχετε χρόνο, ο συνάδελφος μπορεί να σχολιάσει το εμπόριο πολύ σύντομα. Μήπως προτιμάτε να το αναβάλουμε για άλλη φορά για την επόμενη σας συνεδρίαση. Άλλωστε είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτή. Δύο φράσεις μόνο να πω. Καλύτερα να τελειώνουμε με αυτή τη συζήτηση. Τώρα, δύο λεπτά. Σίγουρα το εμπόριο είναι τμήμα της ε, πολιτικής μας, της αναπτυξιακής, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε και χρηματοδότηση. Χθες έγινε μία συνδιάσκεψη υπό την Προεδρία της Εύα Ζολή είναι σημαντικό να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης, ε, γιατί έχουμε πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και καλό θα είναι να τη διαβρύνουμε και με το εμπόριο. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ ζήτησε το λόγο, αλλά παρακαλώ χρόνο φίδου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να αναφέρω μια πτυχή που δεν είχε ακόμα ε, παίξει κανένα ρόλο, αλλά που μακροπρόθεσμα για το θέμα τη χρηματοδότηση για τα συγκεκριμένα θέματα, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Πρόσφατα ήμασταν με την αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη και εκεί η πρόεδρος του ΕΝΤΠ, η Helen Clark, αναφέρθηκε ξεκάθαρα στο ότι τα χρήματα που δίδονται οι ενισχύσει για το, την ανάπτυξη των πόρων κλπ. δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των κλιματολογικών αλλαγών, τη πολιτικής εκεί για αυτό το θέμα και το ανάπαλι, βέβαια. Η χρηματοδότηση δηλαδή δεν θα πρέπει να προέρθει από κεφάλαια που προβλέπονται για την και βοήθεια, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά κονδύλια που θα ε, χρηματοδοτούν από όλα τα κρατη μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Και εδώ πραγματικά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις υποχρεώσεις της στα χρήματα που θα διαθέσει εδώ πραγματικά να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών και η πρόκληση των κλιματολογικών ανάλογων θα πρέπει συμπληρωματικά να χρηματοδοτηθεί. Το λέω αυτό γιατί χθε ελέγχθη ότι το Συμβούλιο Ε, προβλέπει να χρηματοδοτήσει τις στοχότερες χώρες για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών, ε, των συνεπιών μάλλον των κλιματολογικών αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να μην χάνουμε την γενική εικόνα από τα μάτια. Κύριε Higgins, θέλετε να ολοκληρώσετε παρακαλώ. I'll be very brief and then at the end θα είμαι επιγραμματικός και να δούμε και τη συνέχεια. Ο κύριος Μάρτιν αναφέρθηκε στα πνευματικά δικαιώματα τα συναφή με το εμπόριο. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συναφή με εμπόριο. Πολύ σημαντικό. Διατάξεις ε, TRIPS SYN περιλήφθηκαν στην Συμφωνία Οικονομικής Εταιρική Σχέσης με το CARIFORUM αλλά και στην συμφωνία που οριστικοποιείται τώρα με τις ε, χώρες της κοινότητας των άδεων, Κάτι που δείχνει την ε, έλλειψη συνοχής ακριβώς της αναπτυξιακής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τις ε, συνεχιζόμενες συζητήσεις για την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία, εκεί αν εφαρμοστούν τα ποσά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μεταφορά εκατομμυρίων θέσεων απασχόληση προ τη Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα επισημάνουμε για να δείξουμε ποια είναι η στιγμή πραγματικότητα. Αυτά. Καλώς. Αφήνουμε το χρονοδιάγραμμα για αργότερα. Και ολοκληρώνουμε εδώ την τακτική μας συνεδρίαση. So we'll uh, Χωρίς όμως ε, διάλειμμα, περνάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών, που θα γίνει και κλεισμένα των θυρών. Οπότε όσοι δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος αυτήν, παρακαλώ να εκενώσουν την αίθουσα. To Επαναλαμβάνω, η συνεδρίαση από εδώ και